Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της ε, απογευματινής συνεδρίασης. Καλωσορίζω την εξοχότητά του το πρέσβη κύριο κάν Γέγεφ και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να διεξαγάγουμε την ακρόαση για την έκθεση για Κονσάρι με θέμα οι προκλήσεις της εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκή Ένωση Καζαχστάν. Έχουμε μια σειρά εμπειρογνωμόνων. Θυμίζουμε ότι αυτό τον καιρό η Επιτροπή μας με δική της έκθεση εξετάζει τη σύσταση ε, για διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και ε, τη συνεργασία στις 11 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή και τον Νοέμβριο η έκθεση ε, που έχει σχέση με τη διαπραγματευτική εντολή θα ε, ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Γνωρίζουμε ότι στην ακρόαση αυτή θα συζητήσουμε τις δυνατότητες και τις προκλήσεις των σχέσεών μας με το Καζαχστάν που έχουν σχέση όχι μόνο με το εμπόριο και τις επενδύσεις, αλλά και με πολιτικές, ακαδημαϊκές και πολιτισμικές σχέσεις. Επίσης γνωρίζουμε ότι πιο πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, μας ε, κάνουν να ανησυχούμε. Και συνεχίζονται τα προβλήματα σε σχέση με την ελευθερία του τύπου και τις δημοκρατικές αρχές. και γι' αυτό ε, έχουμε την ε, ακρόαση και αργότερα την έκθεση. Πριν δώσω το λόγο λοιπόν στους ομιλητές, θα ήθελα να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονες, αλλά ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μπαρτολότσι που είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας σε Ευρωπαϊκή Ένωση Καζαχστάν, Κυργυζία και Ουσπεκιστάν και για τη σχέση με το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία. Όλα αυτά έχετε τα ολίγα. Ε, να συγκεράσετε λοιπόν αυτές τις χώρες. Παρακαλώ κύριε Μπαρτολότσα έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εξ αρχή να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο Μπρόκ γιατί οργάνωσε αυτό το ε, σημαντικό σεμινάριο στο οποίο όμως δεν θα μπορέσω δυστυχώς να μείνω μέχρι το τέλος γιατί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουμε ψηφοφορίες. Οπωσδήποτε όμως, έστω και για λίγο, έπρεπε, ήθελα να είμαι εδώ ε, σε μια τόσο ενδιαφέρουσα ανταλλαγή ε, απόψεων ε, γιατί πράγματι είναι μια καλή ευκαιρία να ανταλλάξουμε ε, απόψεις για μια χώρα τόσο σημαντική μεγάλη όπως το Καζακστάν. Το Καζακστάν, να θυμίσω εξ αρχή, είναι σημαντικό εταίρο Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικέ και πολιτικέ διμερεί σχέσει αναπτύχθηκαν πάρα πολύ μετά την ανεξαρτησία και οι προοπτικές για περαιτέρω ε, ανάπτυξη των σχέσεων ε, είναι ε, θετικές. Είναι μια χώρα η οποία προήλθε από την Σοβιετική Ένωση και έχει κάνει γιγάντια βήματα προς τα εμπρός τα τελευταία χρόνια. Ως αποτέλεσμα είναι σήμερα μια από τις πιο δυναμικές οικονομίες της περιοχής το επίπεδο ζωής έχει γενικά βελτιωθεί και λόγω των χάρη μάλλον στις ενεργειακές ε, πηγές έχει βελτιωθεί και η οικονομία. Το Καζακστάν εξάλλου παίζει σημαντικό ρόλο σε ολόκληρη την κεντρική ε, Ασία ε, βάσει και των πόρων που προανέφερα και λόγω της ανάπτυξης οικονομίας παίζει πλέον ηγετικό ρόλο στην περιοχή και ε, ε, πλέον εμφανίζεται ως ένα σημαντικός πόλος συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, ε, κατανοεί κανείς άμεσα το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η νέα εταιρική σχέση, οι διαπραγματεύσεις δηλαδή για τη νέα εταιρική σχέση και όσον αφορά ε, το οικονομικό και το πολιτιστικό δυναμικό αυτής της ε, χώρας που μπορεί να προσφέρει πολλά στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε να συμμεριστούμε με τον ε, λαό του Καζακστάν ε, ε, την χιλιετή παράδοση της γνώσης του, την, τις σχέσεις οι οποίες βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην μη προσφυγή σε ένοπλες ή άλλες αντιπαραθέσεις. Βεβαίως παραμένουν προβλήματα. Βεβαίως η χώρα θα πρέπει να κάνει σημαντικές πρόοδους όσον αφορά την δημοκρατική ε, πρόοδο και τον σεβασμό των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι εύκολη η δουλειά αυτή. Τα αποτελέσματα τα οποία έχουν μέχρι τούδε επιτευχθεί είναι βεβαίως θετικά αλλά δεν είναι καθόλου ε, αρκετά ή από μόνα τους ικανοποιητικά. Θα πρέπει να γίνουν βήματα προς τα εμπρός. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση να διευρύνουμε, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας. Τέλος, είμαι πεπισμένος ότι είναι ουσιώδου σημασία να κρατήσουμε μια προσέγγιση ισορροπημένη και συνεκτική και απέναντι στα μεγάλα ζητήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Όντως, μονάχα μέσω του διαλόγου ε, και μέσω της αμοιβαίας ε, συζήτησης και όχι μέσα από αντιθέσεις θα μπορέσουμε να επιτύχουμε όλο και σημαντικότερα αποτελέσματα ακόμα και στον τομέα του εκδημοκρατισμού και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτή την πρόκληση. Θα δουλέψουμε μαζί με το λαό του Καζακστάν έτσι ώστε να να ολοκληρώσουμε την, ε, ε, ε, την διαδικασία εκδημοκρατισμού που έχει ήδη ξεκινήσει και έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πραγματική βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα αυτή. Να συνεργαστούμε, να εργαστούμε μαζί έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές σχέσεις ενισχύοντας τις εμπορικές σχέσεις και κινητροδοτώντας τις επενδύσεις η σχέση μας ε, ε, θα πρέπει να βασίζεται ε, στην αμφίδρομη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό των αρχών, των πολιτιστικών αρχών και της παράδοσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Και έρχομαι τώρα στους εμπειρογνώμονες μας και θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Μαγλέν Λαγουέλ να λάβει το λόγο. Είναι ερευνήτρια στη UCAM και διευθύντρια ε, του προγράμματος της Κεντρικής Ασίας στο Πανεπιστήμιο George Washington. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το δρόμο το τόσο μακρύ να φτάσετε μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρακαλώ να μας ενημερώσετε για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ που με κάλεσατε και που μου δίνετε το λόγο. Ως πρώτη ομιλήτρια θα ήθελα να αναφερθώ στη σχέση μεταξύ ε, ε, του εκδημοκρατισμού και της διακυβέρνησης αφενός και των θεμάτων ασφαλείας αφετέρου. Νομίζω ότι το Καζακστάν πολύ συχνά αποσυνδέει τη δημοκρατική διακυβέρνηση από την ασφάλεια και τίνει να ερμηνεύει την ασφάλεια περισσότερο ε, ως μία απόφυση του Αφγανιστάν ε, αλλά αυτά τα δύο, ε, ο δημοκρατισμός και η ασφάλεια συνδέονται ε, πάρα πολύ και ιδιαίτερα ό,τι αφορά το θέμα της ανθρώπινης ασφαλείας. Η κατάσταση ασφαλείας στο Καζακστάν επιδεινώθηκε σαφέστατα από το 2011 και μετά και έχουμε μία νέα τάση που θα πρέπει να θέσουμε υπόψη των αρχών της χώρας διάφορα θέματα ε, έχουν ενδιαφέρον. Επέλεξα τρία να σας αναφέρω. Το πρώτο είναι η κατάσταση στις φυλακές και στα σοφρονιστικά καταστήματα γενικότερα ε, στο Καζακστάν. Αυτό είναι μια γενικότερη τάση βέβαια, δεν είναι ειδικό το πρόβλημα και ιδιαίτερο στο Καζακστάν και στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα. Στις φυλακές ε, στρατολογούνται και εκπαιδεύονται και εγκληματίες και ε, ακραίοι Ισλαμιστές από διάφορα κινήματα και αυτό ε, είναι μια σοβαρή κατάσταση στο Καζακστάν, ιδιαίτερα σε κάποιες φυλακές ε, επαρχιακές. Ε, και εδώ ανησυχούμε ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις φυλακές ανηλίκων, γιατί οι νέοι τίνουν μέσα στη φυλακή να στρατολογούνται και να ε, έχουν μια προσέγγιση αντικυβερνητική ή ανατρεπτική. Ε, θα πρέπει λοιπόν να γίνουν πιο ε, σοβαρές προσπάθειες κατάρτισης και επαγγελματικής των φυλάκων, των σοφρονιστικών υπαλλήλων. για να ενισχυθεί η ασφάλεια στη χώρα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το όλο δικαστικό σύστημα που είναι σε κακή κατάσταση γενικά και λείπει και η πολιτική βούληση από την πλευρά των Καζάκο για να βελτιωθεί η κατάσταση στη φυλακή. Και ξέρετε υπάρχει και θέμα διαφθοράς στη δικαιοσύνη. θα πρέπει να το συζητήσουμε με τις αρχές του Καζακστάν, να έχουμε ένα διάλογο πιο αποτελεσματικό. Το δεύτερο στοιχείο ασφαλείας που θα ήθελα να αναφέρω αφορά ε, τις ε, υπηρεσίες ασφαλείας και την αστυνομία. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή να δώσει εκεί η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκές αρχές και τα θεσμικά όργανα. Ξέρουμε ότι είναι ευρύτατη η διαφθορά στην Κεντρική Ασία, όχι μόνο στο Καζακστάν και αυτή αντιμετωπίζεται μόνο μετά από τη διεθνή πίεση. Αλλά και αντιμετωπίζεται όταν είναι μεμονωμένοι οι επίουρκοι υπάλληλοι, οι διεφθαρμένοι. Γιατί όταν είναι πυραμίδα και οργανωμένοι είναι πολύ πιο δύσκολο να ε, καταπολεμηθεί. Και η διαφθορά έχει να κάνει κυρίως μεταξύ ανταγωνιστών ε, όταν θέλει κάποιος να... Ε, επικρατήσει. Δεν είναι πρόσφατο το φαινόμενο, αλλά η τάση φάνηκε το 10 και το 11. Όταν έχουμε ένοπλες ε, προστριβές μεταξύ κάποιων συμμοριών ε, και της αστυνομίας, φαίνεται ότι συνδέονται με έναν ανταγωνισμό για τον έλεγχο επιχειρήσεων ή ε, περιουσιών ή στοιχείων ενεργητικού. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί ε, είναι τμήμα της παραοικονομίας που ε, υποτίθεται επισήμως ε, καταπολεμούν και προσπαθούν να πατάξουν. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με τους εταίρους μας εκεί, τις αρχές της χώρας. Και αυτά τα θέματα συνδέονται όλα μεταξύ τους. Ορισμένες υπηρεσίες ασφαλείας έχουν ρόλο στην διακίνηση ανθρώπων, στο δουλεμπόριο κυριολεκτικά και είναι σημαντικό να συνεργαστεί με τις αρχές της χώρας η διεθνής κοινότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαφθορά εντός του συστήματος. Μια αυξανόμενη ανησυχία που συνδέεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας και το θέμα αυτό είναι η έκρηξη των ιδιωτικών υπηρεσιών ε, παροχής ε, ασφάλειας και προστασίας. Ε, security. Είναι ένα θέμα ιδιωτικοποίησης της ασφάλειας και των υπηρεσιών της και ε, το βλέπουμε αυτό και αλλού στον κόσμο, αλλά νομίζω ότι αυτό το στοιχείο πρέπει να ε, ειδωθεί και ε, να προσεχθεί από πολύ κοντά. Γιατί έτσι και η δικαιοσυνική αστυνομία είναι πολύ ασθενής και διεφθαρμένη. Και εκείνοι που δουλεύουν σε ιδιωτικές υπηρεσίες και είναι σωματοφύλακες ε, κάποιων επιχειρηματιών ή προσέχουν τις περιουσίες τους. Είναι πρώην στρατιωτικοί, πρώην μέλη πολιτοφυλακής, πρώην ε, αστυνομικοί και γενικότερα συνδέονται ε, και με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Υπάρχει μια κουλτούρα ατιμορρησίας. και ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος πλήττεται και γενικότερα αυτό είναι βάρος της ασφάλειας στο Καζακστάν και γενικότερα στην περιοχή και σε κάποιες περιφέρειες ε, στη, ε, στη δυτική και στη νότια περιοχή. Ε, τελευταίο θέμα οι θεομηνίες. Ε, και ε, οι βιομηχανικές καταστροφές, περιβαλλοντικές καταστροφές. Προσπαθεί η χώρα, αλλά απέχει πολύ από τη βελτίωση που είδαμε στη Ρωσία σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εκτάκτων ε, Καταστάσεων. Αυτό είναι περίεργο. Η κοινωνία και οι υποδομές της δρούν και αντιδρούν και ο κόσμος ε, εμφανίζει μια ε, δυσφορία και μια ενόχληση γιατί δεν είναι σε θέση η χώρα να αντιμετωπίσει ε, προβλήματα όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες κτλ. Λοιπόν, δεν πρέπει μόνο να καταπολεμηθεί η διαφθορά στα κρατικά όργανα αλλά να ξαναδούν με ποιο τρόπο εξασφαλίζουν την ευημερία και την ασφάλεια των πολιτών. Θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό και στην ευφυΐα. Για την Κεντρική Ασία χρειάζεται και για το Καζακστάν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα είδος αναδιατύπωσης ε, των μυστικών υπηρεσιών. Τι είναι μυστικές υπηρεσίες, τι είναι υπηρεσίες πληροφοριών. Ε, πώς θα τις χρησιμοποιούμε και πώς μπορούν αυτές να δώσουν ευημερία στην κοινωνία. Και οι νέες ε, τεχνολογίες ε, πώς μπορούν να βοηθήσουν στην ασφάλεια μιας χώρας. Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ε, και ελπίζουμε να είναι πιο δημοκρατική η κατεύθυνση που θα πάρει η χώρα για την προστασία του χώρο. Λοιπόν, το Καζαχστάν αντιμετωπίζει προβλήματα που δεν είναι ε, μοναδικά και ιδιαίτερα. Ε, εξισλαμισμός στις φυλακές, ε, ιδιωτικοποίηση των σωμάτων ασφαλείας και των υπηρεσιών ασφαλείας. Αυτά συμβαίνουν και στην Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το περιβάλλον είναι τέτοιο που αυξάνεται ο κίνδυνος στο εσωτερικό της χώρας θα πρέπει οι αρχές ε, του Καζακστάν να καταλάβουν ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση είναι εκείνο που θα τους φέρει στην ασφαλή διακυβέρνηση. Και να έχουμε ένα διάλογο με σημείο πραγματικά κεντρικό ε, τη σχέση της ε, Δημοκρατική διακυβέρνηση με την ασφάλεια. δημοκρατική διακυβέρνηση σημαίνει ασφάλεια, όχι λιγότερη ασφάλεια. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι ε, ευρύτερος και πιο ανθρώπινος ορισμός του τι εστί ασφάλεια και πώς ε, είναι αυτή άρρηκτα συνδεδεμένη με περισσότερη δημοκρατία και καλύτερη διακυβέρνηση του εδώ και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λαριέλε για την παρέμβασή της και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γευγένης Βόχτης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Διεθνούς Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ένωμης Τάξης του Καζακστάν. Παρακαλώ κύριε Ζόφτης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε. Πριν από μερικές μέρες, ε, ο ύποτος αρμοστής ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφερε το Καζακστάν μεταξύ των χωρών που δεν εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως ορθώς κατέδειξε η ύπατη αρμοστία, στο Καζακστάν χρησιμοποιούνται μία σειρά από μέτρα που πηγαίνουν από την απειλή στον εγκλισμό, στο βασανισμό, την, ε, ε, τον εξαναγκασμό κλπ. Για να σας παρουσιάσω ε, σύντομα το θέμα της ελευθερίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν θα πρέπει να αναφέρω εξ αρχής αυτά τα αρνητικά στοιχεία. Τα 15 τελευταία χρόνια δεν έγινε ούτε μια εκλογική αναμέτρηση στη χώρα που να αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΟΑΣΕ η πολιτική αντιπολίτευση δεν εκπροσωπείται στη Βολή. Ένα από τα μεγαλύτερα ε, ο κόμματα της αντιπολίτευσης επανειλημμένα αλλά ανεπιτυχώς τα τελευταία έξι χρόνια προσπαθεί ε, να εγγραφεί στις εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να ε, ενεργήσει σωστά στις πολιτικές του τόπου. Επομένως ε, καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι απλώς ε, τεχνική αλλά ε, ένας τρόπος να μην υπάρξει ελεύθερη έκφραση της βούλησης των πολιτών. Ακόμα ε, και ένας ε, ε, απαγορεύεται το συνεταιρίζεστε, απαγορεύεται η δημιουργία διαδηλώσεων και ακόμα και ένας μόνος του εάν μιλάει θεωρείται συγκέντρωση. Δεν είναι δυνατόν να οργανωθούν διαδηλώσεις ή τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Το 2005 ε, ε, στις, ε, στην, στο Καζακστάν δεν δόθηκε καμία άδεια για οποιαδήποτε διαμαρτυρία και πάντοτε ήταν σταθερή η άρνηση για οποιαδήποτε συζήτηση στην, ε, στο Κοινοβούλιο για όλες αυτές τις διαδικασίες. Ε, ορισμένοι από τους οργανωτές ε, κάποιων εκδηλώσεων μετά το πέρας αυτών συνελήφθησαν και ότι ακόμα και πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδήλωση ή εκδήλωση μπορούν οι συμμετέχοντες ή οι διοργανωτές κυρίως ε, και οι ομιλητές να συλληφθούν ακόμα και πριν ξεκινήσει ε, η διαδικασία. Δεν ε, υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ορισμένα blogs και ορισμένες ιστοσελίδες οι οποίες θεωρούνται αντιπολιτευτικές. Η κατάσταση επίσης των μειονοτήτων είναι πάρα πολύ κακή. Ε, έχουμε μαρτυρίες βασανισμού ιδιαίτερος ε, σε μία από τις αποφάσεις της η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών έχει, έχει αποφανθεί ότι δεν, σημερι δεν συμμορφούνται το Καζακστάν με τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών το Καζακστάν δεν, δεν είναι σε θέση τα, τελευταία χρόνια ε, να αρθεί στο ύψος των διεθνών συμφωνιών και ε, τρεις φορές το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε ότι απεφάνθη μάλλον ε, περί μη του Καζακστάν και το Σεπτέμβριο απεφασίστη η συζήτηση για το ενδεχόμενο επίπληξης προς το Καζακστάν. Ε, γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα ε, δίκη αντιφρονούντος ε, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Χθες ήρθα σε επαφή με τον εκπρόσωπο της Ηνωμένης Ευρώπης υπεύθυνο για τα θέματα του Καζακστάν Συγγνώμη, συγγνώμη. Μήπως μπορείτε, λέει ο πρόεδρος, να μιλάτε λίγο πιο αργά, γιατί δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο για τους διερμηνείς να σας ακολουθήσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεχίζει ο μιλητής, ε, έχει, ε, ε, έχει ήδη ψηφίσει ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στο Καζακστάν. Γνωρίζετε ότι ε, στο Γιανόζιν ε, το, για έναν ε, μήνα είχαμε διαδηλώσεις και απεργίες των εργαζόμενων και των εργατών. Ε, παρόλα αυτά δεν ξεκίνησε διάλογος και περισσότεροι από χίλιοι εργάτες που συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις απελήθησαν. Επίσης, ε, ε, να πούμε ότι ε, αποθήθηκαν οι διαμαρτυρώμενοι και οι συγκεντρωμένοι παρότι δεν είχαν αναλάβει καμία πράξη βίας. Επίσης, ε, οι ειρηνικές, διαδικασίες, οι ειρηνικές διαμαρτυρίες οι οποίες είχαν διοργανωθεί στην ίδια πλατεία που είχαν απεργήσει οι εργάτες ε, των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει μια νέα συγκέντρωση αλλά και αυτή απαγορεύτηκε ε, και σαν αποτέλεσμα της, ε, των, της απόθεσης αστυνομίας είχαμε 15 ε, νεκρούς. Έχει ξεκινήσει υποτίθεται και μια διαδικασία έρευνας όσον αφορά το ε, την ε, ιστορία που σας ανέφερα προηγουμένως. Έχουμε κοινοποιήσει σε όλους, ε, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όλα τα ζητήματα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι μετά το πέρας των δικών, το μόνο που καταφέραμε ήταν να δούμε πολλές καταδίκες εργαζομένων. Πέντε αστυνομικοί πέρασαν από ε, δίκη και στάλησαν όλοι τελικά σε στρατόπεδα εργασίας. Ε, Είναι σημαντικό να υπογραμμίσει κανείς ότι οι αστυνομικοί οι οποίοι ευθύνονται ε, για, τις, ε, για τους θανάτους των εργαζομένων ε, και των διαμαρτυρωμένων τελικά βρέθηκαν στις ίδιες φυλακές με τους εργαζόμενους. Επίσης, σε μια άλλη πόλη του Καζακστάν έχει ξεκινήσει η ποινική δίκη ενός συνδικαλιστή ο οποίος κατηγορείται για υποκίνηση ε, κινημάτων κλπ. Παρακολουθώ την δίκη από την ε, αρχή της. Ε, ο κατηγορούμενος ε, είναι μέλος ενός κόμματος που εδώ και έξι χρόνια προσπαθεί ανεπιτυχώς να εγγραφεί στους καταλόγους, τους πολιτικούς καταλόγους της χώρας. Του αρνείται η κυβέρνηση οποιαδήποτε πρόσβαση στις εκλογικές διαδικασίες. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η εισαγγελία γενικά και τα δικαστήρια χρησιμοποιούν τις παλαιές σοβιετικές μεθόδους. Το ίδιο ισχύει και την ίδια αντιμετώπιση έχουν όλοι όσοι συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς, φόρα, δραστηριότητες κτλ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ότι λαμβανομένων ε, των ε, συνθήκων το πρόβλημα της ε, πολιτικής αντιπολίτευσης όλο ένα και μεγαλώνει, γίνεται πιο δύσκολο και θα δούμε τελικά να αντιμετωπίζουν πρόβλημα όλοι, ακόμα και με μονομένη πολιτικοί αντιφρονούντες υπό το φως των διαπραγματεύσεων που ε, λαμβάνουν χώρα μεταξύ Καζακστάν και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεύρυνση της ε, συνεργασίας ε, σας απευθύνω έκκληση να θέσετε θέμα όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την συμμόρφωση του Καζακστάν προς τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να, και επίσης να σταλούν ανεξάρτητοι ερευνητές για να δουν τι ακριβώς συνέβη στις διάφορες πόλεις τις οποίες ανέφερα προηγουμένως και στις οποίες ε, είχαμε προβλήματα στη διάρκεια ε, διαμαρτυριών. Ε, επίσης να, δούμε, να, να δουν αυτοί οι παρατηρητές τι συμβαίνει με τα μέσα ενημέρωσης και με τα ανεξάρτητα μέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην δόκτωρα Ανδρέα Σμιτ από την Stiftung Wissenschaft und Politik. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σήμερα ενώπιον σας. Ε, σίγουρα το Καζακστάν στην Κεντρική Ασία είναι ο βασικότερος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρεις λόγους βασικά. Πρώτον, το οικονομικό προφίλ της χώρας, ο πλουτοπαραγωγικός της ε, πλούτος ε, και η συμβουλή του στο Διεθνές Καπιταλιστικό Σύστημα και στη συνέχεια είναι εταίρος του ΝΑΤΟ και τρίτον, ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η χώρα για την περιφερειακή σταθερότητα. Εδώ και δύο δεκαετίες δεν υπήρξε κανένα σοβαρό πρόβλημα ε, και θεωρείται ως αξιόπιστος εταίρος των Ευρωπαίων ε, το Καζακστάν και οι, οι δυτικές επιχειρήσεις ευελπιστούν σε προνομιακή μεταχείριση μέσω της σύναψης συμφωνιών με το Καζακστάν. Τώρα, σε σχέση με την πολιτική φιλελευθερωποίηση, τον εκδημοκρατισμό και το σεβασμό του κράτου δικαίου, δεν έχουν υλοποιηθεί οι υποσχέσει ε, του Καζακστάν. Ε ε, φάρο σταθερότητα λοιπόν υπήρξε το Καζακστάν, αλλά αυτό άλλαξε τώρα λόγω διαφόρων ε, συμβάντων ε, που είναι και αλληλένδετα. Ορισμένα αναφέρθηκαν στου προλαλήσαντε. Ε, πρώτον, στο δυτικό Καζακστάν σοβαρέ απεργίε και βίαιη καταστολή το περασμένο Δεκέμβριο. Δεύτερον, Υπήρξαν ε, καταγγελίες ε, για βασανιστήρια που αποσιοποιήθηκαν ε, και δεν γίνεται σεβαστή η σύμβαση του 98 του ΟΗΕ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης φυλακίζονται μέλη της αντιπολίτευσης, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφοι, δικηγόροι για το... επειδή σχολίασαν τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση την κρίση. Ο ύπατος εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα για τα συμβάντα του Δεκεμβρίου ε, σε σχέση με την χρήση βασανιστήριων, αλλά απερίφθη το αίτημα και ο Βλάντιμιρ Κόσλοφ, ο ηγέτης ε, της αντιπολίτευσης, ε, και δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχουν ελάχιστες ε, προϋποθέσεις ε, για το κράτος ε, δικαίου. Αυτό καταδεικνύει ότι χρησιμοποιείται το δίκαιο για πολιτικούς λόγους και ο μοναδικός σκοπός είναι να αποδειχθεί η ενοχή σε μια δίκη. Είναι εντυπωσιακό διότι περισσότερο Όλο και περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν η πολιτική τάξη ε, δεν ε, ε, καταστέλει οποιαδήποτε προσπάθεια να επηρεαστεί επηρεαστούν οι πολιτικές εξελίξεις. Επίσης, σαλαφιστικές ομάδες εμφανίζονται και η οικονομική ευημερία του Καζακστάν δεν εξασφαλίζει την πολιτική σταθερότητα. Τώρα, αυτά τα συμβάντα δεν αποτελούν από μόνα τους ε, τεκμήριο ε, λαϊκής εξέγερσης, όμως ε, δείχνουν δυσαρέσκεια διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη καταστολή της ανεξάρτητης πολιτικής δραστηριότητας και αυτό δείχνει απώλεια της νομιμοποίησης του καθεστώτος και ε, το καθεστώς αυτό όλο ένα ε, και περισσότερο δυσκολεύεται για να ρυθμίσει όλες αυτές τις ασυμμετρίες ε, και τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της κατάστασης. Ε, Ποιε είναι λοιπόν οι προϋποθέσεις για τη σταθερότητα και τι μπορεί να γίνει στο Καζακστάν. Η στρατηγική μας ε, για την περιοχή αυτή βρίσκεται στο πέμπτο έτος υλοποίησης της τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, όχι μόνο στο Καζακστάν αλλά και σε γειτονικέ χώρες. Ε, αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει την δέσμευση ε, ώστε να γίνουν ανοιχτέ κοινωνίες τα κράτη της Κεντρικής Ασίας να προαγάγει τη σωστή διακυβέρνηση και να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών προωθώντας ένα κοινωνικό διάλογο. Αφετέρου όμως πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται στο ότι προβλέπεται σταθερότητα ε, στην περιοχή, υποστήριξη των εκεί καθεστώτων ε, μέσω τεχνολογικής ε, αρρωγής, μέσω αναπτυξιακή βοήθεια. Όμως υπάρχει ταυτόχρονα καταστολή των αντιφρονούντων και απολυταρχικά καθεστώτα όπως αυτό του Προέδρου Ναζαρμπάγεφ καταλαμβάνουν όλο ε, και περισσότερο δημόσιο χώρο όμως ε, αλλάζει η πραγματικότητα ως προς την επικοινωνία και γίνεται ένα και πιο ε, κεντρική διακυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ρηψοκίνδυνο για μας. Δεν μπορούμε να βασιστούμε ε, στη σταθερότητα της περιοχής αν συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίτευξη μόνο των συμφερόντων τους ε, τα πολιταρχικά αυτά καθεστώτα. Θα ήθελα να κάνω και κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις όλων αυτών των παρατηρήσεων που έκανα σε σχέση με την εταιρική σχέση καθώς και τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης. Το Ευρωψήφι ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου 2012 συμπεριλαμβάνει και ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Καζακστάν ε, θα μπορούσαν να αποκομίσουν αμοιβαία ωφέλη από μια βαθύτερη συνεργασία. Όμω ε, η πρόοδο τη διαπραγματεύση ε, για τη Συμφωνία συνήθω πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα ω προ το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Καζακστάν. Πρέπει να καταδειχθεί καλή βούληση του Καζακστάν ναι, να ε, συμμορφώνεται και να προαγάγει τι κοινέ αξίε. αυτή η προπόθεση είναι εκ των όνων κάνεφε για να τελεσφορήσουν οι προσπάθειές μας. Ε, μπορεί να ακούγεται αυτό ε, ω κοινοτυπία, αλλά η διαπραγματεύσεις είναι ένας εύσχημος τρόπος για να κρύψουμε ότι δεν επιδιώκουμε τα σωστά πράγματα. Ποιο συμπέρασμα θα μπορούσα να αντλήσω, το λιγότερο είναι περισσότερο όπως λέμε, δηλαδή ε, ε, ε, αντί θα πρέπει να ορίσουμε προτεραιότητες αντί να προσπαθούμε να καλύψουμε ολόκληρο το πεδίο συνεργασίας. Ε, δεύτερον, χρειάζεται εντατικότερο διάλογος σε σχέση με τα ωφέλη που, στα οποία μπορούμε να προσβλέπουμε με ρελιστικό τρόπο. θα πρέπει να εξετάσουμε διεξοδικότερα το θέμα. Στη συνέχεια, με, ε, αντί να ασχολούμαστε με τα τεχνικά ζητήματα, ε, καλό θα ήταν να βασιζόμαστε, όπως και σε οποιαδήποτε εταιρική σχέση, στις κοινέ μας αξίες. Ε, και η δέσμευση σε σχέση με τις αξίες δεν θα πρέπει να αποδεικνύεται με δηλώσεις, αλλά με απτά και συγκεκριμένα βήματα. Grazie Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Τομπίας Μπάουμαν, υπεύθυνο του τμήματος Ρωσίας Ανατολικής Ευρώπης, Τουρκίας και Δυτικής Ασίας από την Ένωση Επιμελητηρίων της Γερμανίας. Yeah, thank you very much. I would like Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω στα γερμανικά, αν έχω τη δυνατότητα. Βεβαίω, Και όσοι δεν καταλαβαίνετε γερμανικά, παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ έχω υπόψη μου βεβαίως προοπτικές της γερμανικής οικονομίας, αλλά ό,τι θα πω ισχύει γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί καταλαβαίνουμε μετά πώς ανάγεται αυτό στο Καζακστάν και ε, το αντίθετο. Και για την ευρωπαϊκή οικονομία λοιπόν, αλλά και για τη γερμανική οικονομία, το Καζακστάν είναι ο μεγαλύτερος εταίρος και ο σημαντικότερος στην Κεντρική Ασία. Κανονικά δεν φάνηκε αυτό από την αρχή. Η μεγαλύτερη χώρα ήταν το Ουσπεκιστάν με τις καλύτερες προοπτικές, με 25 εκατομμύρια και πλέον κατοίκους. Αλλά το Καζακστάν ε, από την απελευθέρωση της οικονομίας ε, την ανάπτυξη του τομέα των πετρελαίων και ε, του φυσικού αερίου ξεπέρασε το Ουσπεκιστάν τη δεκαετία του 90 και στο μεταξύ το 90 περίπου 100 του εμπορίου με την Κεντρική Ασία δηλαδή με τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες της περιοχής, γίνεται με το Καζακστάν. Οι υπόλοιπες χώρες είναι περιθωριακές μόνο σε αυτή την υπόθεση. Το Καζακστάν είναι μια οικονομία που βασίζεται στις πρώτες ύλες. Το 90 περίπου είναι πετρελοειδή, φυσικό αέριο, προϊόντα ενέργειας και μέταλλα ε, που εξάγονται και στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Η Γερμανία συνολικά στις διμερείς σχέσεις έχει ένα μερίδιο της τάξεως του 25 με 30% αλλά δεν είναι ο πρώτος επενδυτής. Ο πρώτος επενδυτής τα τελευταία χρόνια ήταν οι κάτω χώρες, 40%, η Γαλλία 7,2%, ο Καναδάς και Κίνα ακολουθούν 5 με 6% και η Γερμανία περίπου στην 11η θέση, 1,6% των επενδύσεων. Αυτό τι σημαίνει, ότι το Καζακστάν παραμένει ε, αγορά εξαγωγών ε, ε, για τις εταιρείε της Ευρώπης και όχι τόπος παραγωγής. Ε, αλλά είναι από τις πιο δυναμικές αγορές που έχουμε και που αυξάνεται με το μεγαλύτερο ρυθμό ή από τους μεγαλύτερους. Ετησίως μετά την οικονομική κρίση το ΑΕΠ έχει μια μεγέθυνση κατά 5 με 6%. Οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011 αυξήθηκαν κατά 43%, οι εξαγωγές τους κατά 15% και το διμερές εμπόριο κυμαίνεται ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καζακστάν, δηλαδή ετησίως στα 29 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τη Γερμανία ε, αναλογεί αυτό σε 6,2 δις και κυριαρχούν οι εξαγωγές. Πιο γρήγορα αυξάνονται οι εξαγωγές μας προς το Καζακστάν ε, παρά οι εισαγωγές. 25% ε, αυξήθηκαν πέρσι οι εξαγωγές μας, ενώ οι εισαγωγές κατά 16%. Για να σας δείξω μια τάξη μεγέθους λοιπόν. 6,2 δις από τη Γερμανία και μόνο έχουμε τζίρο, διμερή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σύγκριση με τη Ρωσία 75 δισεκατομμύρια, δηλαδή δεκαπλάσιο και πλέον. Το Καζακστάν, όπως όλες οι χώρες της περιοχής, χαρακτηρίζεται από ε, μεγάλη ανάγκη εξυγχρονισμού και μάλιστα τεχνικού και τεχνολογικού εξυγχρονισμού των διαδικασιών παραγωγής, ε, των υποδομών, ε, των συστημάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, γενικά των συνολικών υποδομών της ιατρικής περίθαλψης των συστημάτων υγείας. Υπό την έννοια αυτή το Καζακστάν ακόμα και αυτό ισχύει, ξέρετε, και για τις υπόλοιπες χώρες κεντρικής Ασίας, είναι ενδιαφέρον ε, τόπος για τις ευρωπαϊκές οικονομίες που το αξιοποιούν αντίστοιχα. Σας είπα από την αρχή ότι ε, ξαναβρίσκει τη ρευστότητα της οικονομίας και τη δυνατότητα να κάνει τον εξυγχρονισμό μετά την κρίση. Ε, ε, αυξήθηκαν και οι τιμές των πρώτων υλών και των καυσίμων. Αλλά είναι πολύ μεγάλη και η εξάρτησή τους από τις τιμές των πρώτων υλών και στις διμερείς σχέσεις ας πούμε η αύξηση που παρατηρείται πολλές φορές συνδέεται και εξαρτάται από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Της τιμής, όχι των ποσοτήτων που διακινούνται. τα ελλείμματα ποια είναι και τα προβλήματα. Ακούσατε και από τους προαλήσαντες. Οι μηχανισμοί λήψη αποφάσεων δεν χαρακτηρίζονται από μεγάλη διαφάνεια ούτε κυβερνητικέ πρακτικές. Είναι μεγάλη η διαπλοκή ε, μεταξύ ε, του δημοσίου και της ιδιωτικής οικονομίας, οπότε αυτό δημιουργεί γραφειοκρατία, εμπόδια, διαφθορά ε, και είναι πολύ λίγη η μικρή παρουσία μικρομεσαίων επιχειρήσεων μεγάλοι τομείς της οικονομίας ε, κατέχονται από μονοπωλιακές δομές ε, με ε, οργάνωση βεβαίως ιδιωτικής οικονομίας αλλά με έλεγχο του κράτους. Παρ' όλα αυτά, γενικά υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες και είναι περισσότερες από τα προβλήματα και τις ελλείψεις. Η στρατηγική βεβαίως της καζακικής κυβέρνησης είναι να ξεφύγει από αυτή την εξάρτηση από τα καύσιμα. Όταν συζητάτε με τους ηθήνοντες εκεί και τους κυβερνώντες σας λέγουν ότι βεβαίως θέλουμε να γίνουμε μέρος παραγωγής ε, βιομηχανικών προϊόντων, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να διαφοροποιήσουμε την οικονομία μας. Αλλά υπολείπεται όμως κατά πολύ ε, το Καζακστάν δεν είναι καθόλου ελκυστική χώρα για επενδύσεις. Θα πρέπει να είναι τέτοιο το πλαίσιο. Πόσο χρόνο έχω? Δεν έχω άλλο χρόνο. Six minutes. I know that. Έχετε άλλα τέσσερα λεπτά. Είσαι στα έξι μόλις. Α, τι έλεγα λοιπόν. Δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για να επιτρέπει ε, αυτές τις επενδυτικές ε, αποφάσεις. Μέχρι τώρα δεν το καταλαβαίνουν πολύ στο Καζακστάν. Θεωρεί ότι ε, είναι ελκυστική η χώρα. Σας είπα για τα καύσιμα. Ε, η τραπεζική κρίση επίσης ε, είναι κάτι που μας απασχολεί. Εάν έχετε ερωτήσεις να απαντήσω στη συνέχεια. α, υπάρχει η Τελωνιακή Ένωση που έχει κάποιες επιπτώσεις και η μελλοντική προσχώρηση του Καζακστάν ε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπόριου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπάουμαν και θα δώσουμε τώρα τον λόγο στον κύριο Γιάπ Δίνεν, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ε, Διεθνής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Παρακαλώ κύριε Βίνεμ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν ο πρόεδρος ε, του Καζακστάν, ο Ναζαρμπάγεφ, παρουσίασε τις ιδέες του για, την κοινωνική, για τον κοινωνικό εξυγχρονισμό του Καζακστάν, με αυτά τα 20 βήματα, ε, αναρωτηθήκαμε αμέσως με ποιους, μαζί με ποιους θα έκανε αυτά τα 20 βήματα. Η Συνομοσπονδία ε, Συνδικάτων, την οποία εκπροσωπώ σήμερα εδώ, δουλεύει με δύο ομοσπονδίες ε, στο ε, Καζακστάν που έχουν ζητήσει να γίνουν μέλη στο ATUC. Είναι πρώτα το FPRK, 2,5 εκατομμύρια συμμετέχοντες παρουσιάζει, έχει περιφερειακές ε, δομές σε όλες τις περιφέρειες ε, και που ε, οργανώνει 38%, συνδικαλίζει 38% των εργαζομένων. Έχουμε και ένα δεύτερο συνδικάτο το οποίο επίσης είναι πολύ δραστήριο. Ε, περιορίζονται τα συνδικάτα ε, στην δράση τους ε, από την περιοριστική πολιτική που ασκούν η κυβέρνηση, που ασκεί η κυβέρνηση αλλά και από τον περιοριστικό εργατικό νόμο ο οποίος δεν κάμπτεται εύκολα οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι και οι ηγέτες του συνδικαλιστικού κινήματος δεν έχουν ε, και εμπειρία ε, όσον αφορά το, τον κοινωνικό διάλογο και από τη φύση τους και λόγω της παράδοσής τους έχουν μεγάλο σεβασμό στους ε, νόμους. Όμως, σε γενικές γραμμές, τα συνδικάτα δεν μπορούν να υπεραμεινθούν ε, τον, σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, έστω και αν έχουν προσυπογράψει και τις 8 συμφωνίες, συνθήκες μάλλον ε, για την εργασία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ε, και έχουν ενστερνιστεί επίσης τις αρχές περί του συνεταιρίζεστε και του οργανώνεστε και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 12 16, Εξακολουθούν ε, να υπάρχουν ε, διαφορές βέβαια όσον αφορά αυτές ε, τις, όσον αφορά τις διαμαρτυρίες οι οποίες οδήγησαν σε θανάτους και σε προβλήματα υγείας το κράτος πάντοτε φαίνεται ότι επιβάλλει μέτρα χωρίς καμία πρώτερη διαβούλευση με τους εργαζόμενους ε, και κάνει όλο και πιο πιεστική την νομοθεσία. Δεύτερον, ε, δεύτερο σημείο είναι ε, το γεγονός ότι τα συμβαλόμενα μέρη δεν έχουν δύναμη. Από τη μία πλευρά τα συνδικάτα ζουν και δρούν σε ένα εχθρικό και ανασφαλές περιβάλλον ε, και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν γίνεται σεβασμό. Ε, η εργοδοσία ε, δεν έχει φερθεί ποτέ καλά δεν προχωράει σε κανονικές διαπραγματεύσεις και ακόμα και οι επενδυτές που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες εταιρείες παραμένουν σιωπηλοί η κυβέρνηση ε, ε, φοβάται ότι εάν ξεκινήσει διάλογο θα ε, ανοίξει την πόρτα για ένα είδος αραβικής άνοιξης. Το 2011 έγινε μια έρευνα από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα πορίσματα της οποίας απολύτως εστερνιζόμαστε τα συνδικαλιστικά κινήματα στο Καζακστάν προσπαθούν να συμμετέχουν, προσπάθησαν μάλλον να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, αλλά έθεσαν τον έλεγχο των διαμαρτυριών ε, και των ε, απεργιών και επομένως ε, πλέον με δυσπιστία τους βλέπουν οι εργαζόμενοι. Η ηγεσία του συνδικαλιστικού κινήματος άργησε να συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται διεθνή στήραξη, συγγνώμη, στήριξη και από την δικιά μας Συνομοσπονδία Συνδικάτων και από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. μαζί με εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας συμπεράναμε ότι η άκαμπτη, ο άκαμπτος και περιοριστικός εργατικός νόμος απαγόρευε στην ουσία την απεργία. Δεν υπάρχει ε, ε, καμία νόμιμη απεργία στα τελευταία 20 χρόνια διακυβέρνησης του Καζακστάν. Ε, υπάρχει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή των συνθήκων ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και αυτή ζήτησε επανειλημμένα από την κυβέρνηση του Καζακστάν να τροποποιήσει τον εργατικό νόμο. Εν τέλει δε, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, εκλήθη να υποβάλει τροπολογίες στο ενεργατικό νόμο του Καζακστάν. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει, βρίσκεται σε εξέλιξη και πολύ πρόσφατα είδαμε ένα προσχέδιο των τροπολογιών αυτών. Αλλά μέχρι τώρα τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Πέρα από τις ε, βελτιώσεις, ε, το προσχέδιο αλλαγών του νόμου προβλέπει ταυτόχρονα ε, πιο αυστηρούς τρόπους λειτουργίας ε, για τα συνδικαλιστικά μέσα ε, και κάνει ακόμα πιο δύσκολη την απεργία την οποία εξακολουθεί να θεωρεί παράνομη ο νόμος και η τάξη σύμφωνα με τις ε, αρχές και την παράδοση του Καζακστάν δεν ταυτίζεται με το πνεύμα των προτινόμενων τροπολογιών ούτε βρίσκει ε, ούτε οι αρχές ε, μπορούν να συμφωνήσουν με τέτοιες τροποποιήσεις μετά από το δράμα και τους ανώσεους υπάρχει ίσως κάποια μικρή ελπίδα ότι η διαδικασία μεταρρύθμισης ε, του συνδικαλιστικού κινήματος του Καζακστάν τουλάχιστον έχει ξεκινήσει. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, και η, Συνομοσπονδία, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία ε, των Συνδικάτων έχει κάνει κάποιες προτάσεις ε, προσπαθώντας να ε, προσέξει περισσότερο την, ε, το συνδικαστικό κίνημα στην περιοχή. Βέβαια ξεκίνησε πολύ αργά αυτή η προσοχή. το διεθνές κίνημα συνδικάτων ε, μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει στείλει πολλές αντιπροσωπείες ε, στο Καζακστάν ε, για να δουλέψουν με τους εργάτες. Και αυτό που είναι σαφές είναι ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κυβερνητική πολιτική ε, νόμου και τάξης και ο τρόπος επιβολής του νόμου οπωσδήποτε θα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να δοθούν ε, κάποιες εξουσίες, κάποιες ελευθερίες στο συνδικαλιστικό κίνημα, τουλάχιστον στις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, για να αλλάξει το κλίμα. πρέπει να πω ότι τα, τον, τον, τα επόμενα χρόνια ε, ίσως να δούμε αυξανόμενη ε, τάση για εργασιακές αντιπαραθέσεις. Βεβαίως τα πρότυπα δημοκρατικά και εργασιακά, έτσι όπως εμείς τα βλέπουμε στην Ευρώπη, σαφώς δεν γίνονται σεβαστά αυτή τη στιγμή στο Καζακστάν. Όσον αφορά την εξέλιξη της εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καζακστάν, βεβαίως εμείς κάνουμε έκκληση για ε, ισχυρές αναφορές ε, οι οποίες θα σχετίζονται με την πλήρη συμμόρφωση προς ε, τις ε, συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που θα τίθενται σε ισχύ, θα υλοποιούνται. Ε, ο εργατικός νόμος, η πολιτική όσον αφορά τις προσλήψεις και τις απολύσεις κτλ. Θέλουμε να είναι δεσμεύσεις που δεν τις αναλαμβάνει μόνο στα χαρτιά η κυβέρνηση, αλλά τις αναλαμβάνει στην ουσία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε τον κύριο Γιάπ ε, Βίνερ για την παρέμβασή του ε, και τώρα θα δώσω τον ε, λόγο αλλά και την Προεδρία γιατί δυστυχώς πρέπει να φύγω να πάω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος γιατί εκεί έχουμε σημαντικές ψηφοφορίες. Δίνω τον λόγο στην κυρία Λίζα Γιακονσάρη, την εισηγήτριά μας. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας που μοιράστηκαν την εμπειρία τους μαζί μας με τόσο ενδιαφέροντα τρόπο. Ακολουθούμε την σωστή κατεύθυνση και είμαστε στο τελικό στάδιο για να καταλήξουμε σε συμφωνία με τους σκιώδεις εισηγητές για τις συμβαστικές ε, τροπολογίες ε, στο ψήφισμα του Μαρτίου, αλλά και τώρα στις συστάσεις μας τονίζουμε ότι η πρόοδος της διαπραγματεύσεις για τη σύνοψη συμφωνίας πρέπει να συνδεθεί με τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις και μια αυθεντική δέσμευση ως προς ε, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον εκδημοκρατισμό. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια των συστάσεών μας. Ζητήσαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, προσφέρει βοήθεια, κατάρτιση, τεχνική αρρωγή για να συμπληρώσει το καλό σχέδιο δράσης ε, του Καζακστάν που όμως ε, δεν ε, χωλαίνει ως προς την υλοποίηση. Όπως μας είπε η κυρία Μαρλένα Λαχιουέλ, υπάρχουν ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφαλείας. Το Καζακστάν θα μπορούσε να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Στο σημείο συνάντησης, ποιο είναι το σημείο συνάντησης όμως της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας, ποιο είναι το σημείο τομής. It's declared Το Καζακστάν θέλει να ακολουθήσει ε, το δρόμο του εκδημοκρατισμού και να τηρήσει τις διεθνείς του ε, δεσμεύσεις. Όμως, υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στους δεδηλωμένους στόχους του σχεδίου δράσης και τις συγκεκριμένες δράσεις. Σε αυτό, σε αυτή σε αυτό τον απολυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης ε, ε, βλέπουμε προβλήματα ε, που ε, δεν μπορούν να επιληθούν και αναρωτιόμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο μεγαλύτερος και ο πλέον αξιόπιστος εμπορικός εταίρος ε, του Καζακστάν με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα το δρόμο της προς τον εξυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό, συγγνώμη, πώς μπορούν να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς μπορούν να δημιουργηθούν συγκεκριμένες ευκαιρίες για τους πολίτες του Καζακστάν ε, και ε, ιδίως ε, για τους νέους. σε μία συνέντευξη στη φιλανδική τηλεόραση με ρώτησαν πιστεύετε, πώς θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 10 χρόνια. Και θα ήθελα κι εγώ να κάνω ένα αντίστοιχο ερώτημα προς τους προσκεκλημένους. Ε, ε ποια θα είναι κατά τη γνώμη σα η θέση του Καζάκσταν ε, στην Κεντρική Ασία σε 10 χρόνια. Πώς ε, προβλέπετε να είναι το μέλλον του Καζακστάν. ίσως περίπλοκο το ερώτημα, αλλά εμένα με απασχολεί. We must have zero tolerance. Για τα βασανιστήρια πρέπει να δείξουμε μηδενική ανοχή. Υπάρχει και μια σχετική μελέτη για τις πιθανές λύσεις, αλλά θα ήθελα εσείς να μας πείτε με ποιο τρόπο θα βοηθήσει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Καζακστάν, ούτως ώστε να μην επαναληφθούν ε, όλα αυτά τα περιστατικά βασανιστήριων. Ποια μέτρα πρέπει να αναλυθούν και πιστεύετε ότι υπάρχει, θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρέσβης ε, στο Καζακστάν έχει έρθει εδώ πέρα και θα σας δώσω το λόγο ενδεχομένως να μπορούσατε να απαντήσετε και σε όλα αυτά τα ερωτήματα που έθεσα. Αλλά ίσως πρέπει να ακούσουμε πρώτα την κυρία Νικολάη από τους ε, φιλελεύθερους. Χαίρομαι που είμαι εδώ, Πρόεδρε, γιατί είναι πολύτιμες οι πληροφορίες ενδιαφέρουσες. Ε, είναι καλή η ε, προσέγγιση όπως σκιαγραφείται από τους ομιλητές. Αλλά ε, όπως είπε ένας από τους ομιλητές, το Καζακστάν είναι εταίρος με λίγα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το γεγονός. Ε, για να έχουμε θετικά αποτελέσματα πρέπει επίσης να ε, καταδείξει καλή βούληση και το Καζακστάν. Ναι. Ε, τώρα, στα συμβάντα τα οποία σχολιάσατε, υπήρξε χρήση βίας, ε, αφέθηκαν ελεύθεροι διάφοροι που είχαν φυλακιστεί μεταξύ των οποίων και εγώ Ε, και κάπως ρυθμίστηκε η κατάσταση αλλά σίγουρα δεν πρέπει να επιτρέψουμε περαιτέρω συλλήψεις ε, πρέπει να φεθούν ελεύθεροι όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί, δημοσιογράφοι όλοι όσοι συνδέονται με την κρίση αυτή Φαίνεται όμως ε, ότι υπάρχει μία ε, κοινή βούληση να είμαστε παρόντες τουλάχιστον να συνεχίσουν το διάλογο και γι' αυτό θα ταχθώ υπέρ των, ε, των διαπραγματεύσεων και φυσικά ε, ευελπιστώ να ολοκληρωθούν. Υπάρχει όμως το πρόγραμμα ε, του Προέδρου Πούτιν για την ολοκλήρωση την ένωση όλων των κρατών της περιοχής ε, και υπάρχει σοβαρός ε, κίνδυνος να υλοποιηθεί. Ξέρω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αρέσει αυτή η ιδέα διότι αν συμβεί κάτι τέτοιο Μπορούμε εμείς να ζητάμε για περισσότερη δημοκρατία, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, σεβασμό του κράτους δικαίου, ε, αλλά δεν θα ωφελήσει σε τίποτα. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την κατάσταση σε σχέση με όλους τους φυλακισμένους, αλλά για να σημειωθεί η επιτυχία δεν πρέπει μόνο να κατακρίνουμε, πρέπει και να δράσουμε. Είμαι υπέρ μιας διερευνητικής αποστολής στο Καζακστάν και θα ε, ε, έπρεπε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υποστήριξη προς την αντιπολίτευση και τους δημοσιογράφους με πολύ συγκεκριμένο όμως τρόπο. Δεν φτάνει να ζητάμε κράτος, δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Πρέπει ειδικά για το, στην περίπτωση του Καζακστάν να αναλάβουμε συγκεκριμένες ε, δράσεις. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νικολάη, που είναι σχεδόν συζητήτρια από πλευρά των φιλελευθέρων, ε, πρέπει να αποχωρήσει και γι' αυτό τη έδωσα ε, πρώτα απ' όλα τον λόγο. Ε, πρέσβη, σας ακούμε. Thank you very much. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, αν δεν έχετε κάποια ένσταση, θα μπορούσα εγώ να παρέμβω μετά το πέρας της συζήτησης. Απάντηση. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κιλ Νίλσεν από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρώ ότι αυτή η ακρόαση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ήταν σημαντικό να διοργανωθεί και είμαι ικανοποιημένη από τις παρεμβάσεις των εμπειρογνωμόνων διότι σκιαγράφησαν ε, ένα πολύ, μια πολύ ενδιαφέρουσα και πλήρη εικόνα της κατάστασης στο Καζακστάν. Ο κύριος Ζόφτης ε, αφέθηκε, αποφυλακίστηκε και είναι παρόν σήμερα και χαίρομαι διότι πολλοί εδώ στο Κοινοβούλιο κινητοποιήθηκαν ε, για την αποφυλάκησή του. Θα θέλαμε να τον χαιρετήσουμε. Να επανέρχομαι τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί φυλακισμένοι, αντιρρησίε, ε, συνήθω αντιφρονούντε ε, στο Καζακστάν και βάσει τη νέα μελέτη ε, του ΟΣΑ και του National Democratic Institute αναφέρονται την δίκη του κυρίου Κόσλοφ. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι με αγγίζει προσωπικά αυτή η δίκη και θα σα εξηγήσω γιατί. Είχα καλέσει τον κύριο Κοσλόφ σε μία ακρόαση που είχα διοργανώσει τον Νοέμβριο του 2011 στο Στρασβούργο. Ο κύριος Κοσλόφ στη δίκη εκείνη Ε, άκουσε τα λεγόμενα του στην ακρόαση του Κοινοβουλίου, παρέθεσαν τις παρεμβάσεις που είχε κάνει δηλαδή το 2011 ε, στο Κοινοβούλιο. Είχαν καταγραφεί οι, παρεμβάσεις του και χρησιμοποιήθηκαν για συκοφαντικούς ε, λόγους ή μάλλον να το πω καλύτερα θεωρήθηκε ότι συκοφαντεί τη χώρα του στο εξωτερικό. Μα είναι σκανδαλώδες και απαράδεκτο. θα πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλάξουμε την ελευθερία έκφρασης. Ε, στο κοινοβουλευτικό μας ε, σώμα ε, ήθιστε να έχουμε ανοιχτές, πολύ ανοιχτές συζητήσεις. Αυτή τη απόδειξη η σημερινή συζήτηση εκπροσωπείται η πρέσβεια του Καζακστάν. Πάρα πολύ ωραία. Όμως, αν η παρουσία των αντιπροσώπων των κρατών έχει τέτοια αποτελέσματα, συλλήψεις δηλαδή, καταγγελίες, κατηγορίες και δίκες, να κάνουμε κάνουμε τις ακροάσεις και κλεισμένων των θύρων. Θα ήταν λυπηρό, γιατί εμείς είμαστε συνηθισμένοι στη διαφάνεια και στο δημοκρατικό διάλογο και είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά για μας, αλλά ε, ε, εφόσον αναφερθήκα συγκεκριμένα στην παρουσία του πρέσβη, ελπίζω να μεταφέρει αυτά που είπα και να τα καταγράψει, όπως έγινε και με τον κύριο Κοσλόφ, ε, και ελπίζουμε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Σε εκείνη την ακρόαση είχαμε και τον κύριο Βινιεύσκη, έναν δημοσιογράφο που επίσης συνελήφθη μετά την ακρόαση. Τώρα αποφυλακίστηκε. Αλλά καν κάθε φορά ε, ε, έχουμε, ακούμε ε, πολύτιμε μαρτυρίε από δημοσιογράφους, από αντιφρονούντες, από οποιονδήποτε και στη συνέχεια φυλακίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Ε, συγγνώμη, τίθεται να αμφιβόλω η ίδια λειτουργία του Κοινοβουλίου. Ε, πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτό συνέβη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Γέγκλε του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, ιδιαίτερα τους πέντε προσκεκλημένους για την ακρόαση. Ε, μας έδωσαν ε, μια ε, ευρεία εικόνα της κατάστασης. Όταν γίνεται λόγος ε, για συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, που ήταν και αφορμή για τη διοργάνωση άλλωστε της ακρόασης, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή η συμφωνία την έχουμε από το 1999. Δεν είναι καινούρια. Μέχρι τώρα έπαιξε σημαντικό ρόλο και τώρα θα πρέπει και οι δύο πλευρές, και το Καζακστάν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, να προχωρήσουν, γιατί θέλουν και οι δύο πλευρές και εμβάθυνση και βελτίωση και διεύρυνση της συμφωνίας αυτής. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ακουστούν και οι δύο πλευρές και να ε, κερδίσουν και οι δύο πλευρές από τη συμφωνία αυτή. Να προχωρήσουμε δηλαδή από κοινού προς την ίδια κατεύθυνση και να είμαστε ισότιμοι ε, και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ακούστηκε ε, από τους προλαλήσαντες και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας δύο πράγματα. Την κοινωνική κατάσταση των πολιτών και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βίνεν που μας παρουσίασε πάρα πολύ ωραία πώς κινούνται τα θέματα και πού παραμένουν προβλήματα. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βίνεν ακριβώς τα συνδικάτα ε, αγωνίζονται για όλους τους εργαζομένους στο Καζακστάν γιατί άκουσα ότι εδώ έχουν προνομιακή θέση οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια. Αλλά εκεί που δουλεύουν αλλού, ε, στη Γεωργία ας πούμε, ε, δεν ε, πρωταγωνιστούν οι εργαζόμενοι. Και οι εργαζόμενοι της χώρας δεν βλέπουν την κατάσταση πάρα πολύ ε, ρόδινη, γιατί λέγουν ότι οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία πετρελαίου κερδίζουν πολύ περισσότερα χρήματα από εμά και γιατί εμείς είμαστε σε μειονεκτική θέση. Λοιπόν, σας ρωτώ, ε, ε, κατανοώ και το αναγνωρίζω ότι στο Καζακστάν υπάρχει και πολιτική βούληση να αλλάξουν τα πράγματα στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα κοινωνικά δικαιώματα και να προαχθούν. Αλλά είναι δύσκολο αυτό. Γιατί είναι δύσκολο, διότι ο κόσμος, οι, πολίτες θέλουν πρώτα απ' όλα σταθερότητα, ασφάλεια και ασφάλεια και επισητιστική για να μπορούν να ζουν στις οικογένειές τους. Η πρόταση που έχουμε ενώπιόν μας και κατέθεση η συγκήτρια, έχουν καταδεθεί και πολλές τροπολογίες, ε, αποτελεί καλή βάση και θα έχουμε τις επόμενες ε, ημέρες και συμβιβασμούς γιατί θα καλέσει συζητήσει που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Για μένα είναι σημαντικό σε μια τέτοια συμφωνία να αναφέρονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καλή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και ο εκδημοκρατισμός αλλά και ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό στα μάτια μου είναι η νεολαία και η εκπαίδευση. Θα πρέπει και εδώ να υποστηρίζουμε και ως ευρωβουλευτές να σκεφτούμε τι κάνουμε εμείς για να ε, δούμε πώς θα προχωρήσει το πρόγραμμα έρεσμος για όλους, γιατί τώρα συζητούμε και τον προπολογισμό των επόμενων ετών. Είναι σημαντική η οικονομία και η κρίση αναφέρθηκε, δεν έχει τελειώσει, πρέπει να γίνουν πολλά σε διάφορες κατευθύνσεις και με το εμπόριο και με το θέμα των επενδύσεων. Το Καζακστάν δεν είναι σημαντική χώρα μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ενεργειακά, είναι κομβική χώρα στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας και για την ενέργεια και για το περιβάλλον και για τη διαχείριση των υδάτων και για τις μεταφορές αλλά και για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και την ε, ασφάλεια των συνόρων. Ε, από εκεί που περνάνε τα ναρκωτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα βεβαίως και την ασφάλεια των ανθρώπων. Αλλά θα πρέπει ε, να κερδίσουν και οι δύο πλευρές από τη συμφωνία αυτή. Νομίζω αυτή η προθυμία είναι δεδομένη από πλευράς μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μέρφυ της ΓΚΟΕ. Ε, σας ευχαριστώ ε, ε, για τις παρουσιάσεις σας. Ενημερωθήκαμε όπως πρέπει για το τι συμβαίνει στο Καζακστάν. Οι διαπραγματεύσεις για την σύναψη συμφωνίας είναι εξαιρετική ευκαιρία τους ώστε να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει επί τόπου, κυρίως σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατικά δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα και νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε σε αυτά που συμφώνησε το Κοινοβούλιο το Μάρτιο, δηλαδή ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων διαπραγματεύσεων θα πρέπει να είναι συνάρτηση της προόδου των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω καμία πρόθεση να επιβάλλω σε οποιονδήποτε ευρωπαϊκές ε, αξίες. Συχνά η κυβέρνηση του Καζακστάν ε, ε, αντιπροτάσει αυτό το επιχείρημα ότι προσπαθούμε να επιβάλλουμε τις αξίες μας. Όταν πήγα στο Καζακστάν το αίτημα για πραγματικά δημοκρατικά δικαιώματα, ελευθερία του συνέχεια, έρχεστε, η ελευθερία της έκφρασης κτλ. Όλα αυτά τα αιτήματα προέρχονται από ε, τους πολίτες, από τους γεωργούς, από τους εργαζόμενους και ε, προ ε, και σίγουρα δεν έρχονται από το εξωτερικό. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει σημαντικές επιλογές. Ε, τα εμπορικά της ε, συμφέροντα καθώς και τα πολιτικά και γεωπολιτικά της συμφέροντα τελικά υπερσκελίζουν αυτή την απλή δήλωση για την προστασία του, κρατού, κράτους δικαίου, των εργασιακών δικαιωμάτων κτλ. Και γι' αυτό τονίζω ότι είναι σημαντικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι χάρη σε αυτό μπορούν να ενωθούν οι δύο εργατικές ε, τάξεις, ε, η ευρωπαϊκή ε, και η καζάκικη και να σημειωθεί μία πρόοδος. Και από αυτή την άποψη μπορούμε να εξετάσουμε το αν ήδη έχει σημειωθεί πρόοδο. Ε, κατά τη γνώμη μου δεν έχει σημειωθεί πρόοδο τον τελευταίο χρόνο και αυτό προκύπτει και από την έκθεση. Μάλλον το αντίθετο καρκινοβατή το Καζακστάν ε, στο Τζένοζεν η σφαγή που έγινε συνιστά καμπή ε, οι, οι εργαζόμενοι καταδικάστηκαν σε, όπως και οι αξιωματούχοι της αστυνομίας. Έγιναν πολλές καταγγελίες για βασανιστήρια. Στη συνέχεια ε, χρησιμοποιήθηκε αυτή η κρίση για να γίνουν επιθέσεις ε, κατά της Ε, Είδαμε τι έγινε με την δίκη του ε, κυρίου Κοσλόφ. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται σε αυτές τις δίκες, η ηχογράφηση, η, όπως είπε η κυρία Κιλ Νίλσεν, οι τηλεφωνικές υποκλοπές εναντίον των ακτιβιστών ή οποιονδήποτε μαρτύρων, τα προβλήματα μετάφρασης, δεν δίνεται χρόνο χρόνος ε, ε, για να εξεταστεί και να εμπεδοθεί το υλικό της δίκης. Το Φεβρουάριο άλλαξε και το ποινικό δίκαιο στην χώρα ε, και νομιμοποιήθηκαν οι απολύσεις των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις όταν κάνουν παράνομες απεργίες. και Ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε ε, τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο ευρωπαϊκής συνεργασίας. Δηλαδή, ε, στην Ιταλία μεταξύ άλλων άρχισε μία δίκη κατά τη CNI που είναι μία πετρελαϊκή εταιρεία που και δεν είναι η μόνη, υπάρχουν και γερμανικές, ολλανδικές που δέχονται κατηγορίες για διαφθορά για τις επιχειρήσεις τους επιτόπου στο Καζακστάν. Σα ε, ε, σας ευχαριστώ, αλλά είναι λίγο περιορισμένος ο χρόνος μας, ε, λέει η Πρόεδρος, ο κύριος Ρούσεκ και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον πρέσβη και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα και σε εσά να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Παρακαλώ. E e Αναφέρθηκε ότι το 2010 έγινε μέλος του ΟΣΕ βλέποντας ε, και τη διαδικασία αυτή και τη διαδικασία του Ελσίνκη τη δεκαετία του 90 θα ε, δούμε ότι υπάρχουν τρία καλάθια. Το ένα ε, ήταν πολιτικό στρατηγικό, το άλλο οικονομικό, εμπόριο, οικονομικές ανταλλαγές και τρίτο ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικά δικαιώματα. Ε, στα πλαίσια αυτά τη ε, διαδικασία αυτής δηλαδή η Δύση δούλεψε μαζί με την Ανατολή και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό και αν δεν ήταν καλό ε, δεν θα ήμουν και εγώ σήμερα καθισμένο εδώ γιατί έρχομαι από πρώην κομμουνιστική χώρα. ο ΣΑ και η, ο ΑΣΕ και οι αρχές του είναι το σωστό όχημα για να συνδυαστούν αυτά τα τρία στοιχεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως και επομένως ε, και το Καζακστάν και όλη η Κεντρική Ασία ε, θέλουμε να έχουν πολιτική σταθερότητα και βεβαίως και εκείνη το ίδιο και ε, θέλουμε και τις εμπορικές συναλλαγές, φυσικά και εκείνοι το θέλουν, αλλά και εμείς θέλουμε να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζομένων κλπ χωρίς καταστολή από κυβερνήσεις αυταρχικές ε, ή τουλάχιστον να βρούμε κάποια ισορροπία μεταξύ των τριών αυτών ε, πόλων, των τριών επιπέδων που ανέφερα προηγουμένως. Αλλά από την άλλη πλευρά είμαστε πολιτικοί και ξέρουμε ότι όλα αυτά, όλη αυτή η διαδικασία δηλαδή δεν ε, γίνονται σε κενό, δεν λαμβάνουν χώρα σε κενό. υπάρχουν χώρες μεταξύ ε, ημών και το Καζακστάν, υπάρχει ας πούμε η Ρωσία. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα ε, να ρωτήσω πώς βλέπουν τα όσα λαμβάνουν χώρα στη Ρωσία τώρα και βεβαίως ε, και βεβαίως ε, ε, τι λένε οι Ρώσοι, τι λένε οι κάτοικοι του Καζακστάν όσον αφορά την Ευρωασιατική ε, Ένωση. Θέλουν την Τελωνιακή Ένωση, θέλουν άλλου είδους ένωση, γιατί και αυτό θα έχει αντίκτυπο στις σχέσεις που θα έχουμε με το Καζακστάν. Η ερώτησή μου... Απευθύνεται στους πανελίστες λοιπόν τι αντίκτυπο θα έχει η ευρωασιατική ένωση που θέλουν και οι ηγέτες του Κρεμλίνου και οι ηγέτες του Καζακστάν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ, σύντομα παρακαλώ, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, ήθελα απλώς να καταγραφεί ότι η ομάδα των ε, συντηρητικών, ε, θέλει ισχυρέ σχέσει με το Καζακστάν, ε, να έχει δηλαδή ευρωπαϊκή σχέση, σχέσεις με το Καζακστάν. Όταν πρώτο ήρθα σε αυτή την επιτροπή ήμουν από αυτούς που στα πλαίσια της ανατολικής πολιτικής γειτονίας ζήτησα, επέμεινα να μπει και το Καζακστάν. Είναι γείτονα της Ευρώπης το ε, ε, Καζακστάν και μάλιστα έχει για ένα τμήμα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι ε, είναι δίπλα στην Ευρωζώνη. Ε, έχει το καλό να συνδυάζει μουσουλμάνους με χριστιανούς ε, και αυτοί οι πληθυσμοί να ζουν ε, σε ηρεμία και ειρήνη μεταξύ τους. Επίσης είναι σημαντική σύμμαχη στην καταπολέμηση της τροποκρατίας και του θρησκευτικού ριζοσπαστισμού. Και από την άλλη πλευρά είναι πηγές, είναι χώρα με μεγάλες δυνατότητες όσον αφορά πρώτες ύλες, ε, πετρέλαιο, αέριο, ουράνιο κτλ. Ε, και ε, και βεβαίω εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε το Καζακστάν να ευθυγραμμιστεί μόνο με τη Ρωσία ή με την, ε, ε, με την Κίνα. Είναι γεγονός και το δέχομαι ότι βρίσκονται σε, ένα μεταβατικό δημοκρατικό στάδιο. έχει υπάρξει επιλεκτική δικαιοσύνη, υπάρχουν οπωσδήποτε υπάρξει και ομότητες και ε, βίαιες καταστολές. Είμαι ο πρώτος που θα το πει. Ε, και αυτά μας διαφοροποιούν, διαφοροποιούν το Καζακστάν από την Δύση. Ε, από την ε, άλλη πλευρά νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν και μία μακρά παράδοση μουσουλμανικών πληθυσμών, έχουν μία μακρά παράδοση όσον αφορά... So, thank ε, σοφών και άρα και από αυτό θα πρέπει να μάθουμε κι εμείς. Ευχαριστώ. Ε, ξέρετε, εμείς στο Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, δεν μιλάμε πολύ συχνά πάνω από δύο λεπτά ο καθένας Είναι μεγάλη πολυτέλεια, λοιπόν, που μπορείτε να ε, μιλήσετε. Κύριε ε, Πρέσβη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι αυτή η ακρόαση που ετοίμασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούσαμε σήμερα μια ευρεία έτσι, έποψη στοιχείων ως νεοδιοριστής πρέσβης του Καζακστάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπω ε, την ε, ε, αποστολή μου να μεταφέρω τα στοιχεία αυτά στην κυβέρνησή μου και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είμαι ανοιχτό προς όλους, προς όλους τους μετέχοντες στο ακροτήριο αυτό και στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στους ομιλητές που είναι εμπειρογνώμενος ο καθένας στον τομέα του και μας είπαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εδώ σήμερα. Επίσης είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε μορφή συζήτησης, ανταλλαγή απόψεων, ε, που θα αφορά είτε τους στόχους, τους σκοπούς της κυβέρνησης είτε τις θέσεις της κυβέρνησης. Ξέρετε πολύ καλά ότι η χώρα έχει ξεκινήσει την οδό του εξυγχρονισμού. Ξέρετε ότι η χώρα βρίσκεται ε, σε μεταβατική περίοδο ε, και από άποψη οικονομική και κοινωνική και πολιτική βλέπουμε την ε, ανάπτυξή μας, την εξέλιξή μας ως δυναμική δομή. διαπιστώνουμε την μεγάλη σημασία των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ επιβεβαιώνω εδώ την πολιτική βούληση που έχει η χώρα μου ε, για διαπραγματεύσεις ε, με ειρηνικό και επικοδομητικό τρόπο έτσι ώστε να είναι ε, αμφιδρόμως αποφελές το αποτέλεσμα και η έκβαση αυτών των συνομιλιών. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ε, ε, Συμφωνία εταιρική Σχέσης. Θα πρέπει να δουλέψουμε μαζί. έτσι ώστε και το Καζακστάν να γίνει αξιόπιστος εταίρος και χώρα σημαντική στην Κεντρική Ασία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστούμε και καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες, λοιπόν, λέει η κυρία Γιακονσάρη. Θα δώσω τώρα το λόγο στους καλεσμένους ομιλητές ε, και πρώτα απ' όλα στον κύριο Γιάπ Βίνεν. Για πολύ λίγο, δύο λεπτάκια κύριε Βίνεν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 40% των εργαζόμενων του Καζακστάν είναι ε, συνδικαλισμένοι στα συνδικαλιστικά κινήματα τα οποία συνεργάζονται μαζί μας. Έρχονται δε από όλες τις ε, ε, ομάδες εργαζομένων. Η, ε, η Διεθνής Συνομοσπονδία γνωρίζει τις ε, συνδικάτων, γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες και αυτό που θέλουμε εμείς ε, είναι και τα συνδικάτα στο Καζαστάν ε, να ακολουθούν τις δικές μας αρχές, δηλαδή ακεραιότητα και ανεξαρτησία. Βεβαίως οργανώνουν ε, τα συνδικαλιστικά τους κινήματα με τον τρόπο που εκείνοι επιλέγουν. Δεν μπορούμε να σας αποβάλουμε εμείς κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπάουμαν, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια μόνο να πω για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα δύο για την Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμπόριο μόνο με χώρες που είναι ε, δημοκρατικές και έχουν τη δική μας αίσθηση και αντίληψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν το ζήτησε κανείς αυτό, άλλωστε είναι και ένα εδαφικό. Αλλά η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων φέρνει ένα νέο πολιτισμό, μια κουλτούρα στις χώρες αυτές και χρειάζεται κάποιο χρόνο για να ευδοκιμήσει και να προχωρήσουν στον εκδημοκρατισμό και στη μεγαλύτερη διαφάνεια. Ε, να είναι αυτό υποστηρικτικό, ας πούμε, των θετικότερων εξελίξεων. Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές μας σχέσεις. Αυτές συνδέονται με κατάρτιση, με εκπαίδευση, με κατάρτιση εργαζομένων και είμαστε βέβαιοι ότι ε, συνεισφέρουμε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Για την ευρασιατική οικονομική κοινότητα νομίζω είναι σαφές. Η Ρωσία φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα οικονομικό συνασπισμό εκεί, όπου να ελέγχει την περιφέρεια. σχετικά. Η ίδια. Είδαμε με την Τελωνιακή Ένωση ότι οι χώρες που συμμετέχουν, Λευκορωσία και Καζακστάν, έχουν αναλάβει κατά 86% να ε, μεταφέρουν ε, ό,τι ίσχυε ε, για τις τελωνιακές ρυθμίσεις της Ρωσίας, χωρίς να έχει απαραίτητος πλεονεκτήματα για τις χώρες αυτές κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή στους θεσμούς, ας πούμε, η κοινότητα κρατών και ε, πώς θα μεταξελιχθεί και τι θα κάνουν και χώρες μεταξύ τους σε σχέση με τις διάφορες ε, υποθέσεις πολιτικές και οικονομικές. Ε, νομίζω είναι πολύ νωρίς για να έχουμε τώρα οριστική άποψη γι' αυτό. Ευχαριστώ ε, η κυρία Ανδρέα Σμιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρία σημεία μου επιτρέπετε. Σύντομα θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση που κάνατε εσείς στην αρχή. Πώς βλέπουμε το Καζακστάν σε δέκα χρόνια. Ε, ποιες θα είναι οι τάσεις τότε, οι σημερινές που οδηγούν προς τα εκεί. Φοβούμε ότι εάν οι σημερινές πολιτικές τάσεις επικρατήσουν στο Καζακστάν, σε δέκα χρόνια θα έχουμε ένα κράτος αυταρχικό τάξης ε, και νόμου, πολύ λιγότερο φιλελεύθερο από το σημερινό. Δεν θα είναι βέβαια προς το συμφέρον μας αυτό, πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε. Ε, σε ό,τι αφορά την πρόταση ε, που έγινε, να δούμε το Καζακστάν ως ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, αμφιβάλλω αν αυτό αποτελέσει κίνητρο για την πολιτική ηγεσία του Καζακστάν. Είδαμε με την προεδρία του ε, ε οπισθοδρόμησε όλα στη χώρα τον καιρό που προέδρευε στον ΟΑΣΕ. Είναι μεγάλα και ωραία τα λόγια και μεγαλεπίβολα τα σχέδια, αλλά στην πράξη δεν γίνεται τίποτα. Και αφιβάλλω εάν αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνητρο, επαναλαμβάνω, για να έρθει το Κασαχστάν ε, στο δρόμο που επιθυμούμε. Ανταυτού θα πρότεινα να παραμένουμε σε αυτή τη ρίση που λέει ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες δηλαδή. Είναι πάρα πολύ αναγκαίο να να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην κοινωνία, να βλέπουμε και πώς ελέγχονται ε, ε, πολιτικά πράγματα, τα πολιτικά σκάνδαλα, ε, πώς μεθοδεύονται κάποιες πολιτικές δίκες. Δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να μην εμπλεκόμαστε, ας πούμε, και να μπούμε σε αυτή την επιχειρηματολογία των ίσων αποστάσεων ή της σχετικής απόστασης δεν είναι θέμα αρχών και αξιών, αλλά ότι ε, η κυβέρνηση του Καζακστάν έχει δεσμευτεί η ίδια τουλάχιστον στα χαρτιά για κάποιες αρχές και αξίες. Ας μην διστάσουμε λοιπόν καμία φορά να συγκρουστούμε κιόλα. Ευχαριστώ. Ο Γευγένη Σόφτης. Ευχαριστώ. Ένα σύντομο σχόλιο. Εγώ πιστεύω ότι αν η κυβέρνηση Ε, καταστέλει και καταπατά ε, μια, καταπατά μια ειρηνική αντιπολίτευση ε, μέτριοπαθή και συγκρατημένη, δημιουργεί ένα κενό το οποίο κενό θα έρθουν να καλύψουν οι ακραίοι εξτρεμιστές ομάδες και απόψεις τους που βλέπουμε σήμερα να αναδύονται στο Καζακστάν. Και όταν φύγουν και από το Αφγανιστάν οι συμμαχικές δυνάμεις θα είναι ακόμα πιο σοβαρή αυτή η απειλή. Δεν είναι μόνο το θέμα της δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Ακόμα σημαντικότερη είναι η ασφάλεια. Θα πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση ε, κοσμική, λαϊκή, ε, μετριοπαθής, ανθρώπινα δικαιώματα, ε, ελεύθερος τύπος, γιατί αυτή είναι η εγγύηση. Δεν μπορεί να πατάσετε τόσο βία και να καταστέλλετε αυτή η μετριοπαθής αντιπολίτευση. Δεν θα λυθούν έτσι τα θέματα, θα έρθουν οι ακραίοι μετά. Ευχαριστώ. Thank you and... Uh, Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρλέν Λαρουέλ, παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα. Το μικρόφωνο, παρακαλώ. Yeah, very briefly on the question of the role of Europe in uh, security για το ρόλο της Ευρώπης σε θέματα ασφαλείας θα πρέπει να αρνηθούμε, να απορρίψουμε αυτά που λέει η κυβέρνηση του Καζακστάν, ότι ε, το πρόβλημα της ασφάλειας ε, απλώς έχει μεταφερθεί από το Αφγανιστάν, είναι το τράφικινγκ, τα ναρκωτικά και τα λοιπά, ότι είναι εισαγόμενο το πρόβλημα. Όχι θα πρέπει η Ευρώπη να ανταπαντήσει με μια άλλη αφήγηση ας πούμε. Να πούμε ότι στο εσωτερικό της χώρας θα πρέπει να δημιουργηθεί ασφάλεια, να υπάρχει πραγματική ε, διακυβέρνηση και σε θέματα ασφαλείας και να ζητήσουμε βελτίωση και διαφάνεια στη διακυβέρνηση των κρατικών οργάνων που είναι επιφορτισμένα με θέματα ασφαλείας. Αλλιώς ε, τα επόμενα χρόνια διακυβεύεται η ίδια η ασφάλεια της χώρας και η σταθερότητά της. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση αυτή. Θα, θα συζητήσετε και με τους βουλευτές και τους συναδέλφους. Ε, θα δείτε και τα ψηφίσματά μας και είναι πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαμε για την έκθεσή μας. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Καζακστάν ανοίγει μεγάλες δυνατότητες η συνεργασία, αλλά αντιμετωπίζει και μεγάλες προκλήσεις όπως ακούσαμε. Τέλος, θα ήθελα όλους ιδιαίτερως να ευχαριστήσω ε, τη Διεθνή Εταιρική Σχέση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που ε, επέτρεψε τη διεξαγωγή αυτή της ε, ακρόασης και ευχαριστούμε και τον Πρόεδρο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον κύριο Σόφτης. Ε, ζητώ συγγνώμη, ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας, αλλά σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Με πρωτοβουλία της ηγήτρας κυρίας Όγιου Λαντ, Έχουμε τώρα μια συζήτηση για την έκθεση της, μάλλον σύσταση προς το Συμβούλιο, σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων έναντι αξιωματούχων της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Μαγνίτσκι ή που ευθύνονται για αυτήν. Δεν είναι καινούρια αυτή η ιστορία. Ε, πολλά κοινοβούλια και στην Ένωση και παγκοσμίω έχουν ασχοληθεί με το θέμα και απεφάνθησαν υπέρ περιορισμών ταξιδίων και μέχρι και για πάγωμα ε, των περιοσιακών στοιχείων Ρώσων αξιωματούχων ε, που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση του κυρίου Μαγνίτσκι. Το συζητάει αυτή τον καιρό και το Αμερικανικό Κογκρέσο και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η υπόθεση δείχνει πώς χρησιμοποιούν στη Ρωσία το δίκαιο για πολιτικούς σκοπούς. Έγινε και συζήτηση, θα θυμάστε την περασμένη εβδομάδα, στο Κοινοβούλιο και υπάρχουν θέσεις που μας ε, καλούν ε, να δραστηριοποιηθούμε σχετικά. Είναι εδώ ο κύριος Πλάουντερ, ε, επικεφαλής ε, της οργάνωσης που αγωνίστηκε υπέρ του κυρίου Μαγνίτσι, ο οποίος εργαζόταν στην εταιρεία του. Και η ίδια η εταιρεία γνωρίζει δυσκολίες ακριβώς. Αυτό ε, είναι μια ιστορία ε, παλιά. Ε, Επισκέφτηκαν τα γραφεία της εταιρείας εκπρόσωποι του Υπουργείου Εστερικών. Της Ρωσίας δεν το συζητούμε για πρώτη φορά το θέμα και προτείνω να ακούσουμε τον κύριο Πράουντερ, τον διευθυντή της εταιρείας, 5-6-7 λεπτά, τον καλωσορίζω θερμότατα και μετά τους κοιόδης ηγητές των πολιτικών ομάδων. Θα πρέπει να τους δώσουμε και την ευκαιρία να ακούσουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης για να μας δώσουν ε, συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε. Στα έγγραφά σας έχετε και το αντίστοιχα έγγραφα της προτάσεις ε, του Κοινοβουλίου και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε και τον ε, Μιχαήλ Κασιάνοφ, πρώην Πρωθυπουργό της Ρωσίας. Καλώς όρισες, Μιχαήλ. Και ε, θα ήθελα τώρα αμέσως να δώσω το λόγο στον κύριο Πράουντερ. Um, <clears throat> uh, Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή ευκαιρία να μιλήσω ενώπιον σας. Ε, δεν είναι η πρώτη φορά. Ε, που έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχω έρθει επανειλημμένα για να συζητήσουμε για την υπόθεση Μαγνίτσκι. Νομίζω ότι πολλοί γνωρίζετε ε, τις περισσότερες λεπτομέρειες της υπόθεσης. Ε, σήμερα θα ήθελα να σας πω τι θα κάνουμε σε σχέση με τις δράσεις των Ρώσων και θα αναφερθώ σε κάποια στοιχεία μιας παρουσίασης που είναι σε μια μελέτη, μια, οθόνη πίσω μου. Πριν από τρία χρόνια περίπου πέθανε υποκράτηση ο Σεργέη Μαγνίτσκι ε, ξέρουμε ότι την τελευταία νύχτα ξυλοκοπήθηκε άγρια και υπάρχουν και αυτές αποδείξεις φωτογραφίες που βλέπετε ε, και αυτό, αυτή ήταν και η αιτία θανάτου βασανίστηκε όσο καιρό ήταν υποκράτηση και έχουμε και άλλες αποδείξεις. Είναι η καλύτερα τεκμηριωμένη υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία τα τελευταία 25 χρόνια κατά πάσα πιθανότητα και είναι καλά τεκμηριωμένη γιατί ο ίδιος ε, έγραψε 450 καταγγελίες, 58 ημέρες παρέμεινε υποκράτηση. Ε, ξέρουμε ποιος ε, του έκανε τι, ε, έχουμε υπογραφές για την ε, ψευδή σύλληψη, παραδείγματο χάρη, για να μην του χορηγηθεί η ιατρική περίθαλψη συγγνώμη, όταν το χρειαζόταν. Ε, οι Ρώσοι είναι υπεύθυνοι, έχουμε τα ονόματα των υπευθυνών, όμως ε, από τους 60 υπεύθυνου που προετοίμασε η Επιτροπή ΙΠΑ Ελσίνκη, που συγκροτήθηκε για το, να ερευνήσει το θάνατο, έχουν απαλλαγεί όλοι εκτό από έναν ιατρό που βρίσκεται στο κατώτερο επίπεδο ε, και ε, για αμέλεια, για επιμελή διάγνωση ε, κατηγορήθηκε και όχι για την άρνηση να παράσχει ιατρική περίθαλψη που είναι ο ουσιαστικός λόγος. Υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις, πάρα πολλές δίκες στη Ρωσία που έχουν γίνει για αυτό το θέμα, αλλά έχουν όλοι απαλλαγή. Και σκεφτήκαμε, ωραία, τι είναι αυτό τώρα και τι να κάνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό το έγκλημα δεν είναι θρησκευτικού χαρακτήρα, ιδεολογικού χαρακτήρα, ε, είναι καθαρά οικονομικό έγκλημα. Ο κ. Μαγνίτσκι αποκάλυψε την εμπλοκή διαφόρων κυβερνητικών αξιωματούχων ε, που έπαιξαν ένα ρόλο για την κλοπή 230 εκατομμυρίων από την ρωσική κυβέρνηση, εξού και η ψευδή σύλληψη, τα βασανιστήρια, αρνήθηκε να δώσει ψευδή μαρτυρία και έτσι ε, δολοφονήθηκε. Πρόκειται για οικονομικό έγκλημα δεν βρούμε την, ε, το δίκαιο μας ε, στη Ρωσία, σκεφτήκαμε πώς αλλιώς μπορεί να γίνει αυτό. Βρήκαμε και τα χρήματα. Ο, ε, Ο ταγμαρτάρχης ε, Κάρποβ έχει καταχραστεί 1,3 εκατομμύρια ε, και έχει ένα μισθό 7.200 ε, δολάρια το χρόνο έχοντας όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Στη συνέχεια του Κουτζνέτσιοφ που ήταν ο αξιωματούχος ο οποίος έδωσε την εντολή για την σύλληψη ε, ε, του ε, ε, βγάζει 10.200 το χρόνο ενώ η οικογένειά του έχει 3 εκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία. Η κυρία Δε που έδωσε την έγκριση για την έκνομη φορολογική επιστροφή έχει ετήσιο μισθό 38.381 και τα περιουσιακά της στοιχεία πλησιάζουν το εκατομμύριο. Ο Ελβε Ελβετικό Γενικό Εισαγγελέα αποφάσισε να παγώσει ένα μέρο αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Πρόσφατα κάναμε καταγγελίε σε 7 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ε, εμφανίστηκαν ε, τμήματα αυτών των ποσών. Ε, στη συνέχεια ανακαλύψαμε ότι δεν πρόκειται μόνο για τα 230 εκατομμύρια που εκλάπησαν, αλλά μετά το φόνο του κυρίου Μαγνίτσκι ε, εκλάπησαν και άλλα 370 εκατομμύρια μετά τη δολοφονία του. Τους αρέσουν τα λεφτά. Ε, και τους αρέσουν και τα ταξίδια επίσης. Ε, έχουμε όλο το ιστορικό τους και βλέπουμε εκατοντάδες ταξίδια, μεταξύ των οποίων και ταξίδια προς την Ευρώπη. Λοιπόν, αν δεν μπορούμε να βρούμε το δίκιο μας ε, στη Ρωσία, τι μπορούμε να κάνουμε εκτός, αναρωτιόμαστε. Αν τους αρέσουν τόσα λεφτά και θέλουν να τα ταξιδεύουν και να τα ε, δαπανούν στην Ευρώπη, ας μην, ας μην τους το επιτρέψουμε. Ε, ε, ήταν πολύ ενεργό το Κοινοβούλιο για αυτή την υπόθεση. Τρία ψηφίσματα υπάρχουν. Δεκέμβριο 2010, 2011 και Μάιο 2012 ε, που όπου καλούμε για, ε, καπευθύνουμε ε, έκκληση μάλλον για πάγωμα περιουσιακών στοιχείων από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Μέχρι στιγμή όμω δεν έχει γίνει τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκανε αυτέ τι ε, κλήσει και ταυτόχρονα άλλε χώρε και άλλοι διεθνεί οργανισμοί ενεπλάκησαν. ΕΙΠΑ, Καναδά, Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη και διάφοροι άλλοι. Επιπροσθέτως, ε, σε αυτές τις ε, κοινοβουλευτικές εκκλήσεις, ε, αν θέλετε. Έχουμε ε, σύσσωμη την αντιπολίτευση, ο Πρωθυπουργός Κασιάνοφ, παραδείγματος χάρη, κάνει αντίστοιχες εκκλήσεις. Ήταν πρωθυπουργό ο κ. Κασιάνοφ και όχι υπουργό παρά το πρωθυπουργό. Υπάρχει λάθο στη διαφάνεια. Συνοψίζοντα, τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα έπρεπε να συντάξει ένα κατάλογο αξιωματούχων που ευθύνονται για τη δολοφονία και την κάλυψη της δολοφονίας στη συνέχεια ε, καθώς και για την παρενόχληση, τη διαρκή παρενόχληση της οικογένειάς του μετά τη δολοφονία πρέπει να απαγορευτούν τα ταξίδια του στην Ευρώπη, να παγώσουν τα περιουσιακά τους ε, στοιχεία για εκείνους και για τους άμεσους συγγενείς τους ε, σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει και πάλι να απευθύνουν επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις προς τη Ρωσία για τη διεξαγωγή έρευνας, αλλά όχι μόνο για τον Σιγκέι Μαγνίτσκι, αλλά και για τις υπόλοιπες τα υπόλοιπα υπέσχυντα εγκλήματα που συμβαίνουν στην Ρωσία. Εκατοντάδες τέτοιες υποθέσεις υπάρχουν με πολύ λίγες διαφορές ε, και εγώ ε, γυρνάω γύρω-γύρω και προσπαθώ να κάνω κάποια πράγματα, τουλάχιστον να σώσω τις ζωές μελλοντικά κάποιων άλλων που θα βρεθούν στην ίδια θέση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πράουτα. Το λόγο έχει τώρα η συγγήτρια μας, η κυρία Ογιουλάντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να προσθέσω κάτι σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Μπράουντερ. Θα ήθελα ε, να σας πω ότι σε 7 παρατέταρτο στην αίθουσα ASP 5G1 ε, θα προβληθεί μια ταινία. Ελπίζω να σας ε, ε, έχουν απευθυνθεί οι προσκλήσεις και να τις λάβατε όλοι εγκαίρως. Σε ό,τι αφορά την έκθεση, αυτή τη σύσταση μάλλον καλύτερα, θέλω να σας πω το εξή Ότι από τον Ιούλιο που συζήτησε για πρώτη φορά την έκθεση επιτροπή μας, έχουμε ακούσει απόψεις διαφόρων πολιτικών ομάδων και μέχρι τώρα είχα μια σειρά ε, συζητήσεων ε, με τους συναδέλφους, πολύ επικοδομητικών και καρποφών 11 τροπολογίες κατατέθηκα για το σχέδιο ψηφίσματος και οι περισσότερες για μένα ως εισηγήτρια ε, είναι αποδεκτές. Σε δύο τροπολογίες έχω ένα ερωτηματικό δεν μπόρεσα να δεχτώ την τροπολογία επαριθμών 10 για τον εξής λόγο. Πρώτον είναι γλωσσική, επαναλαμβάνει το πρώτο τμήμα της ίδιας παραγράφου, αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος, δεν μπορώ να τη δεχτώ διότι θα μπορούσε ενδεχομένως να περιορίσει τις δράσεις των κρατών μελών και των κυβερνήσεών τους όταν θα δεήσουν να πάρουν αποφάσεις για τους περιορισμούς ή το πάγωμα ε, των περιοσιακών στοιχείων. Επίσης, το συζήτησα με τον κύριο Προτασίεβιτς που είναι ο συντάκτης τροπολογίας και του είπα είτε να την αποσύρει είτε θα απορριφθεί ε, γιατί δεν μπορώ να την υποστηρίξω. Και έχω και ένα δεύτερο θέμα να σας αναφέρω. Αφορά τροπολογία 11, είναι ίσονο σημασία αυτό, αλλά εκεί συμφωνήσαμε με τον κύριο Προτασίεβης, γιατί και αυτή είναι δική του, να αποσύρει μία λέξη από την τροπολογία του, ε, που είναι, λέει εδώ, των κοινών βασικών αξιών, shared. Δεν νομίζω ότι έχουμε κοινέ αξίες Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία. Αυτή τη στιγμή καθόλου. Και ε, κατά τα άλλα ε, η τροπολογία είναι εντάξει. Αν βγει η λέξη αυτή κοινών αξιών, κοινών βασικών αξιών. Εμπλουτίζει η τροπολογία αυτή τη σύσταση και θυμίζει τη Ρωσία τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Προτασίεβιτς. Που είναι και από το Βρότσλαβ. Thank you, ε, Ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με τις παρατηρήσεις που έκανε η κυρία Όγιουλαντ, ναι, σε, να συζητήσουμε τις τροπολογίες. Θα συζητήσουμε λοιπόν αυτή που είναι πιο εύκολη να την εξηγήσω. Δηλαδή, την τροπολογία 11. Εγώ πρότεινα τη λέξη ε, shared values, κοινών αξιών, με την έννοια ότι ε, υπάρχουν κοινέ αξίες τις οποίες συμμερίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία. Βεβαίως εδώ σε αυτή την έκθεση μιλάμε για αξίες οι οποίες προφανώς δεν είναι κοινέ, αλλά αναφέρομαι γενικά ε, στην ιδέα των κοινών βασικών αξιών. Γι' αυτό λέω και όπως το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, βασική ελευθερία κτλ. Βεβαίως μπορώ να κατανοήσω ότι ενδεχομένως μπορεί να παρεξηγηθεί αυτή η έννοια. Γι' αυτό λοιπόν ε, εγώ ή το ΕΛΚ δεν θα έχουμε πρόβλημα να υπερψηφίσουμε ε, την τροπολογία της κυρίας Όγιουλαντ, δηλαδή να ε, διαγραφεί η λέξη shared στα αγγλικά, κοινών αξιών στα ελληνικά. Όσον αφορά τώρα την ανθρωπολογία. Το συζητήσαμε και στην προπαρασκευαστική μας ε, συνεδρίαση. Αναμφίβολα ε, η υπόθεση Μακνίτσκι είναι αυτή που είναι. Και δεν ε, λέω ότι δεν δέχομαι ότι υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Όμως τέτοιου είδους διπλωματικές κυρώσεις όπως είναι η απαγόρευση θεώρησης ταξιδίου, βίζας. Ε, πρέπει να θεωρούνται το τελευταίο βήμα, η τελευταία καταφυγική, όχι η πρώτη. Και αυτό δεν είναι μόνο ε, δικιά μου γνώμη, είναι και άλλων ε, μελών του ΕΛΚ. Η τροπολογία αυτή δείχνει ότι βεβαίως ενθαρρύνουμε το Συμβούλιο να ε, ε, τηρήσει την ίδια στάση και σε άλλες περιπτώσεις παρόμοιες. Αλλά ότι τέτοιου είδους μέτρα, όπως είναι η απαγόρευση βίζας, ε, θα πρέπει να είναι το έσχατο μέτρο. Και ευελπιστούμε βεβαίως ότι τέτοια προβλήματα θα μπορούν να λυθούν με την ρωσική πλευρά με πιο διπλωματικό τρόπο ε, ή πιο ευρωπαϊκό αν θέλετε τρόπο. Χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να προσφύγουμε σε αυτά τα έσχατα μέτρα τα οποία είναι διπλωματικά και είναι πολύ βαριά. Όμως συμφωνήσαμε να κάνουμε μια τροποποίηση. Δική μας ε, πρόταση, όχι της κυρίας Όγιουλαντ αντί να πούμε βάση, ε, ότι ε, λέει ας πούμε, ως έσχατο μέτρο υπό τον όρο ότι υπάρχει σαφής απόδειξη του αδικήματος ή της διάπραξης εγκλήματος. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι, το, ότι ε, ο επιθετικός προσδημός σαφής ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Σαφής αποδείξεις ίσως είναι υπερβολικό. Δεν είμαστε και πολύ τόσο αφελείς. Γι' αυτό λοιπόν, εάν ε, μπορούμε να πούμε ε, convincing evidence, πιστικές αποδείξεις που μπορεί να έρχονται από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, από οπουδήποτε αλλού, αυτό μας αρκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο, μπορεί βάσει αυτών των πιστικών αποδεικτικών στοιχείων να πάρει την απόφαση. Επομένως, συμφωνούμε να ε, διαγράψουμε τη λέξη ε, στην τροπολογία 11, στην ΕΔΕ τροπολογία 12, αντί να πούμε «σαφής απόδειξη», να πούμε ότι υπάρχει πιστική απόδειξη, «convincing evidence». Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σάλα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ και η πολιτική μου ομάδα, η πολιτική ομάδα των σοσιαλιστών δηλαδή, μπορεί να συμφωνήσει με την εισηγητρία. Νομίζω ότι η υπόθεση του Σεργέη Μαγνιτσκή είναι ε, μια, ε, ένα ε, παράδειγμα παράφορης καταβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα για λόγους οικονομικούς όπως μας είπε ο κύριος Μπρόντερ προηγουμένως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει πραγματικά να ε, λάβει υπόψη του το ενδεχόμενο της απαγόρευσης ε, παροχής ε, βίζας καθώς επίσης και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων και των οικογενειών τους. Γιατί αυτό είναι και σύμφωνα με την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει της ε, έκθεσης Watson για το θέμα. Δηλαδή, η χρήση των στοχευμένων ε, κυρώσεων, εφαρμογή λοιπόν στοχευμένων κυρώσεων σαν ένα νέο εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα χωρίς όμως να δημιουργήσει γενικευμένο πρόβλημα στην ε, κοινωνία της χώρας προς την οποία η κύρωση απευθύνεται. βεβαίω εμεί μπορούμε να στηρίξουμε και άλλε τροπολογίε που έχουν υποβληθεί στην έκθεση αυτή. Δεχόμαστε όλες τις τροπολογίες οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υπόθεση Μαγκνίσκη. Νομίζω ότι είναι καλογραμμένη, απτή και συγκεντρωμένη η έκθεση και επομένως θα ζητήσω από την πολιτική μου ομάδα να στηρίξει το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέει ο Σούλτς. Οι τροπολογίες μας που είναι συμπληρωματικές και διευκρινιστικές γίνονται δεκτές από την εισηγήτρια, οπότε εγώ δεν θα ε, επεκταθώ ούτε θα ε, μακρηγορήσω. Θέλω να επικεντρωθώ στο πολιτικό ε, ζήτημα που μας απασχολεί εδώ και καιρό και δεν είναι μονομένη τραγική περίπτωση όπως προσπάθησε να την παρουσιάσει πρόσφατα ο κύριος Πούτιν. Είναι κατάφορη και κραυγαλαία περίπτωση και πολύ καλά τεκμηριωμένη. Ο θάνατος του Σεργέη Μαγνίτσκι δείχνει πώς ε, η αυθαιρεσία στη δικαιοσύνη και η διαφθορά στο κράτος ε, μπορεί να οδηγήσει σε τέτοια φαινόμενα και μέχρι τη δολοφονία. Γιατί η ρωσική πλευρά υποσχέθηκε ε, ότι θα το διερευνήσει και θα ξαναέξει την υπόθεση, αλλά αυτή η υπόθεση τραβάει εδώ και χρόνια. Και έχει έρθει η ώρα εμείς να πάρουμε μια στάση ε, στεναρή, αποφασιστική, δηλαδή να πούμε ότι δεν αφήνουμε εγκληματίες να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, αξιοποιούν τους λογαριασμούς τους και να ε, έχουν διάφορες δραστηριότητες και θα πρέπει αυτό να αφορά και τα παιδιά τους. Και δεν θα πρέπει να ε, έχουμε φόβους και αγωνίες γιατί η υπηρεσία εξωτερική δράση φοβάται τα αντίπεινα. Αυτό είναι μια ε, καινή απειλή ότι δεν θα αφήσουν, λέει, υπαλλήλου Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, ταξιδεύουν. Στην Ευρωπαϊκή ε, Γραφειοκρατία, στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση δεν υπάρχουν διεφθαρμένοι εγκληματίε. Τι είναι αυτά Σήμερα ε, περνάει με ρυθμούς ε, βιομηχανικής παραγωγής η Ρωσική ε, Δούμα καταπιεστικούς και κατασταλτικούς νόμους, ε, τροχάδιν. Και δεν θα πρέπει εμείς να δεχτούμε αυτά και να επιτρέψουμε αυτές τις αυθαιρεσίες. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ. Υποστηρίζει η πολιτική μου ομάδα το ψήφισμα της κυρίας Ογιουλάντα και δράτω με τι ευκαιρίε ε, για να χαιρετήσω και, και ε, τον κύριο Μπράουντερ και να, να το αποδώσω τα εύσημα γιατί αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι τη ζωή τα τελευταία χρόνια για αυτήν την υπόθεση για να επικρατήσει δικαιοσύνη και αν δεν ήταν εκείνος ε, και το αξιέπαινο έργο του δεν θα είχαμε ούτε αυτό το ψήφισμα. Ε, αντίστοιχα ψηφίσματα έχουμε από την Βρετανική Βουλή. Νομίζω ότι πρόκειται για στοχευμένες ε, κυρώσεις ε, και ε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της ήπιας εξουσίας που μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιες υποθέσεις. Την περασμένη εβδομάδα συζητούσαμε ένα ζήτημα για το Αζερβαϊτζάν για πολιτικές δολοφονίες. Ε, συζητήσαμε το θέμα των πολιτικών κρατουμένων στην Ουκρανία. Παραδείγματος χάρη η Γιούλια Τιμοσέγκο με ε, ολόκληρος ο χώρος ε, που διαδέχθηκε την Σοβιετική Ένωση έχει παρεμφερεί προβλήματα εκδημοκρατισμού, κράτους δικαίου και διεφθαρμένοι ολιγάρχες διοικούν αυτές τις χώρες και ακολουθούν μια διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή. Πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν χώρες όπως η Ρωσία μπορούν να παραμείνουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης υποτίθεται ότι βασίζεται στο κράτος δικαίου και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία αυτό το θεσμικό όργανο. Ε, για το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο το ίδιο. Είναι λίγο παράδοξο να χρειαστεί να επιβάλλουμε κυρώσεις ε, για θέματα βασικά όπως ε, επιβολή του νόμου και κράτους δικαίου ε, στη Ρωσία. Εγώ θαυμάζω αυτό το κράτος αλλά απορώ που παραμένει μέσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Γεννώνται διάφορα ερωτήματα ερωτηματικά και ε, μήπως θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την περίπτωση ως ε, μια προσωμείωση για να δούμε σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο σε σχέση με την Ρωσία, πώς ακριβώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους κυρώσεις, τέτοιου είδους μέσα. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι υποστηρίζουμε και τις τροπολογίες καθώς και τη διαγραφή του όρου share, ε, δηλαδή δεν είμαι και πολύ σίγουρο τα πόσα μοιραζόμαστε τελικά από πλευράς αξιών και τα λοιπά με τη Ρωσία. Ο κύριος Λαντσμπέργκερ. Πρόεδρε, καλό είναι το ψήφισμα, όσο και απαραίτητο. γιατί αυξάνονται τα προβλήματα στη δικαιοσύνη της χώρας αυτής. Κοιτώ όμως τη τελευταία διατύπωση ε, της τροπολογίας 10 και την παράγραφο αυτή. Νομίζω ότι είναι κακώς διατυπωμένη. Πρώτα, έχουμε δύο όρους που συνδέουμε με τα μέτρα. Πρώτα λέει βάση καλά τεκμηριωμένων. Τι θα πει καλά τεκμηριωμένα στοιχεία. Δεν μου αρέσει αυτό. Λες και απολογούμαστε και ζητούμε συγγνώμη δύο φορές. Α, συγγνώμη για τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλουμε. Γιατί δηλαδή δυο φορές να ζητάμε συγγνώμη. Και ε, ότι να είναι τα, τα έσχατα μέτρα, ως έσχατο μέτρο. Και αν δεν είναι αποτελεσματικό το έσχατο μέτρο, υπό την κυριαρχία του κυρίου Πούτιν, γιατί να πούμε ότι αυτό είναι το έσχατο μέτρο και μετά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Να πούμε κατάλληλο μέτρο ενδεδειγμένο, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το σαφές και το φυσιολογικό. Και τώρα ξανακοιτάω αυτό το σχέδιο και λέει να θεσπίσει περιοριστικά μέτρα ως έσκατο μέτρο. Καλά, ποιος το έγραψε αυτό, κανένας αναλφάβητος. Και γιατί μπορεί να μας εκθέσει εμά ολόκληρο το κοινοβούλιο να ψηφίσουμε ένα τέτοιο πράγμα. Πώς να το χαρακτηρίσω κιόλας. Είναι φτωχό το κείμενο. Εγώ προτιμώ το αρχικό. Και αν υποστηρίξουν οι φιλελεύθεροι το αρχικό κείμενο, ας αφήσουμε τους σοσιαλιστές να απομονωθούν. Αυτά, τελείωσα. Next ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Σεργέη Μαγνίτσχη δολοφονήθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 2009. Στην ετήσια μας έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Δεκέμβριο του 2010 τη σχετική σύσταση. Εγώ ήμουν εισηγήτρια και υπάρχει μία παράγραφος που αναφέρεται σε αυτή την υπόθεση συγκεκριμένα ε, και καλούμε τις δροσικές αρχές ε, να διερευνήσουν κατά το δέον ε, την υπόθεση και να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι και θεωρήθηκε ότι προσπαθούμε εμείς να επιβάλλουμε τη θέλησή μας. Ε, προτείναμε και πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων. Έχουν περάσει δύο χρόνια έκτοτε. Ε, φτάνει, αρκεί. Ε, ε δεν χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να διερευνηθεί σωστά μια υπόθεση και να κινηθούν δικαστικέ διαδικασίε. Ε, υποστηρίζω το σχέδιο ψηφίσματο τη Κριστίνα Ογιουλάντε και προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία. Είμαι πρόθυμη να την υποστηρίξω. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κάλιν. Κέλαν. Ευχαριστώ. Αργήσαμε με αυτό το ψήφισμα υπερβολικά και ευχαριστούμε την συνάδελφο Γιουλάντε που συνέταξε το ψήφισμα διότι δεν πρόκειται τόσο για τη Ρωσία και τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, πρόκειται για την ίδια την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι μέχρι του δε οτιδήποτε και να συμβαίνει στη Ρωσική Ομοσπονδία, τι κάνουμε εμείς, αυτοπεριοριζόμαστε σε εκφράσεις του τύπου ανησυχούμε τονίζουμε την ανάγκη να ε, ε, διορθωθεί η κατάσταση. Αν δεν είμαστε έτοιμοι να ε, επιβάλλουμε πόνο στην Ρωσία μέσω κυρώσεων δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Είναι χρυσή ευκαιρία διότι ε, οι Ρώσοι αξιωματούχοι, οι ίδιοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ε, Ρωσία, ε, στη ρωσική κυβέρνηση και επενδύουν τα χρήματά του στην Ευρώπη. Αλλά άσχετο αυτό. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμά μα δεν πρέπει να δείχνει δισταγμό. Πρέπει να ε, δράσουμε ομόφωνα και να υποστηρίζουμε τις ίδιες ε, αξίες ε, για, τις οποίες, για την προστασία των οποίων έχει δεσμευθεί και η ίδια η Ρωσία. Μόνο έτσι θα βοηθήσουμε τους πολίτες, ε, την κοινωνία των πολιτών, αλλά και εν τέλει την κυβέρνηση της Ρωσίας για να αλλάξει επιτέλους προς το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε. Ε, κυρία Τάραντ, είναι η επόμενη ομιλήτρη, ο κύριος Τάραντ, συγγνώμη, είναι ο επόμενος ομιλητής. Υποστηρίζουμε το ψήφισμα. Έχω όμως μια ερώτηση προς την εισηγήτρια. Θεωρητικό ερώτημα θα θέσω. Αναμένετε να λάβουμε να λάβουμε σύντομα ένα κατάλογο ή περιμένετε ότι θα δείξουν ότι κινητοποιούνται αλλά τελικά δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Και δεύτερο ερώτημα. Πιστεύετε ότι αυτός ο κατάλογος θα συνάδει με τον κατάλογο που μας έδωσε ο κύριος Μπράουντερ ή περιμένετε να κατονομαστούν και υψηλό, ε, πιο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι που ευθύνονται για την δημιουργία ε, αυτού του συστήματος ε, και όχι μόνο για την εκτέλεση των διαταγών στα πλαίσια αυτού του καθεστώτος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζάλα, τελευταίος ομιλητής, παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ. Μία παρατήρηση, μία διευκρίνηση θα ζητήσω σε σχέση με την παρατήρηση του κυρίου Λαντσμπέργκης. Δεν πρόκειται για ένα εργαστήρι των σοσιαλιστών για αυτό το έσχατο μέτρο. Ο κύριος Προτασίεβιτς από το ΕΛΚ υπέβαλε την τροπολογία. Έτσι για να ξεκαθαρίζουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πούλκα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Τέσσερι παρατηρήσεις θα κάνω. Πρώτον, η σύσταση του ΕΛΚΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγγνώμη, είναι θεμητή και ε, ενσωματώνεται σε ένα συνολικότερο πλαίσιο της τάσης δηλαδή του Κοινοβουλίου ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για αυτό το ζήτημα και φαίνεται ε, η σημασία που προσδίδει η Ένωση σε αυτή και σε άλλες τέτοιες υποθέσεις. Επίσης νομιμοποιεί την συνεχή άσκηση πίεσης προς την Ρωσική Ομοσπονδία ούτως ώστε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεύτερον, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την ύπατη εκπρόσωπο συνεχίζουν να απευθύνουν εκκλήσεις προς τη Ρωσία για να διεξαχθεί ε, ιδέουσα έρευνα. Έχουμε μετέλθει όλων των ε, δυνατών μέσων ε, και έχουμε συζητήσει το θέμα σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στο ύπατο. Εσχάτως θέσαμε και το ζήτημα στις 20 Ιουλίου στις διαβουλεύσεις που κάναμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα θυμάστε ότι όταν η ύπατη εκπρόσωπος απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά ε, με το θέμα του δικαστικού συστήματος στη Ρωσία αναφέρθηκε αυτό το ζήτημα τον Απρίλιο το 2012 ο κύριος Ρομπή απέστειλε επιστολή στον τότε πρόεδρο Μετβέτχευ ε, ε, όπου ζητούσε συγκεκριμένη πρόοδο στην υπόθεση Μαγνίτσχη και εκεί σε αυτή την επιστολή απίφθινε τρία συγκεκριμένα αιτήματα. Πρώτον, ε, να ολοκληρωθεί η έρευνα ε, να ε, κλείσει η υπόθεση δίωξης του κυρίου Μαγνίτσχη και τρίτον να να σταματήσουν διαδικασίες για την σύλληψη της μητέρας του και άλλων μελών της οικογένειας του και ε, και θα ήθελα τώρα να σχολιάσω το για ποιο λόγο τα κάνουμε όλα αυτά. Για τρεις καλούς λόγους. Ο πρώτον είναι η φύση της υπόθεσης που μας την παρουσίασε σήμερα ο κύριος Μπράουντερ με ε, ε, ιδιαίτερη παρησία και πρόκειται για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέτοιες υποθέσεις είναι αντίθετες με τις βασικές αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η Ρωσία έχει ίδια συμφέρον να επιλύσει αυτή την ε, υπόθεση που είναι χαρακτηριστική για την κατάσταση ε, του δικαστικού συστήματος ε, στη χώρα αυτή και ε, επίσης τίθεται ζήτημα αξιοπιστίας που είναι σημαντικό και για τις επενδύσεις και για τις επιχειρήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν εκεί για να γνωρίζουν σε ποιο πεδίο, σε ποιο πλαίσιο αναπτύσσουν εκεί τις δραστηριότητες πολίτες τους. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε συμφέρον να είναι σταθερή, βιώσιμη η Ρωσία και να υπάρχει ένα κρατεό ε, κράτος δικαίου στα ε, σύνορά μας Είδαμε ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από ρωσικής πλευράς. Παραδείγματο χάρη είδαμε ένα περιορισμένο άνοιγμα σε, από πλευράς ρωσικής κυβέρνησης. Φωνασκούσε συχνά ο κ. Μετβέτχεφ για την υπόθεση αυτή. και έκτοτε, ε, μάλλον και δεν είχε γίνει ανεξάρτητη έρευνα. Ο κύριος Πούτιν τώρα στην πρώτη επίσημη συνέντευξή του αναφέρθηκε σε αυτό το συμβάν και μίλησε για την ανάγκη να προχωρήσει η υπόθεση. Τώρα βεβαίως πέρα από τις ε, δηλώσεις ε, θα αναμένουμε συγκεκριμένη δράση από ρωσικής πλευράς και φτάνω στο τελευταίο μου σημείο. Τι έπεται εξετάζουμε επιμελώς τις συστάσεις του Κοινοβουλίου καθώς και τα μέτρα που προέρχονται ε, από τις ΗΠΑ. Τονίζω ότι Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η χρήση των ακυρώσεων ε, είναι διαφορετική στις ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου είναι διαφορετικό και το πολιτικό τοπίο. Όπως είπαν και άλλοι, τα περιοριστικά μέτρα είναι ένα ευαίσθητο εργαλείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και ε, δυνάμει των κατευθυντηρίων γραμμών που εμείς έχουμε θέσει. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται ως έσχατο μέτρο ε, και προϋποθέτει το ύψιστο δυνατό επίπεδο πολιτικής υποστήριξης ε, από τις πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας αυτό κατά νου πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση που ε, ασκούμε και έχει συσσωρευτεί για αυτήν και άλλες ε, παρεμφερείς υποθέσεις, ε, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει επίσης να ε, εγγράψουμε αυτή την υπόθεση σε ένα γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή το κοινωνικοπολιτικό πεδίο στην Ρωσική Ομοσπονδία, κάτι που μας ανησυχεί και έχουμε συζητήσει ε, επανειλημμένα και σε σχέση με τα μέτρα που ήδη έχουν αναλυφθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Miss Christina Oyuland. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κριστίνα Όγιουλαντ. Ναι, πριν όμως ε, φτάσω συμπεράσματα θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πούλτς. Μία επιπλέον ερώτηση σε σχέση και με αυτό που ρώτησε ο κύριος Τάραντζα. Ε, δηλαδή, τι θα κάνει συγκεκριμένα και απτά η υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πάρει γιατί νομίζω ότι στην ουσία δεν ανταποκρίνεται στις παρούσες δραστηριότητες και στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτά που ακούσαμε μόλις δεν ε, προσθέτουν οτιδήποτε στα υφιστάμενα μέτρα και στις δυνατότητες τις οποίες έχουμε ασκήσει μέχρι τώρα. Ε, ε, βεβαίως εμείς περιμένουμε και ποιοτικά μια διαφοροποίηση γιατί τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να ξέρουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Θα θέλαμε να μας πει ο κύριος Πούλης ποια είναι αυτά τα επόμενα βήματα ε, και ε, να μας πει ακριβώς τι προτίθεται η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να κάνει. Ευχαριστώ. Yes, if, Θέλετε να απαντήσετε. Θέλετε να απαντήσετε. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Όπως είπα και προηγουμένως, βεβαίως θα μελετήσουμε πολύ προσεκτικά τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν αυτές θα εγκριθούν και υπό το φως αυτών των συστάσεων θα δούμε ποια είναι τα βήματα, τα περαιτέρω βήματα τα οποία θα πάρουμε και βεβαίως θα λάβουμε υπόψη μας και τα υφιστάμενα εργαλεία. Δεν μπορώ τώρα να κάνω οποιασδήποτε ε, σκέψεις ή να προδικάσω οποιασδήποτε πολιτικές αποφάσεις. Τούτη τη στιγμή τουλάχιστον δεν μπορώ να το κάνω. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε αύριο για το θέμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, Δύο λόγια εν συμπεράσματι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που δούλεψαν για το θέμα αυτό και που εξακολουθούν να δουλεύουν. Και να απαντήσω σύντομα στην ερώτηση του κύριου Τάρανς που βεβαίως είναι πολύ σημαντική. Ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία <clears throat> πρέπει να πάρουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων να εγκριθεί γρήγορα στην Ολομέλεια ε, το ζήτημα αυτό και να μην παραμείνει σε ένα σερτάρι. οι πολιτικές ε, ε, ομάδες είναι ενωμένε σε αυτό. Σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πολλά εργαλεία στην διάθεσή μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τους συναδέλφους μας στα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι να διατηρήσουμε την πίεση προς τις εθνικές κυβερνήσεις και στρέφομαι προς όλους σας έτσι ώστε να συνεργαστούμε μεταξύ μας και να συνεργαστούμε και με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο θέμα είναι η κατάσταση στη Συρία. Και καλωσορίζω τον κύριο Ιγμιν Γενικό Διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Αραβική Χερσόνησο, το Ιράν, το Ιράκ. Α, ε, ε, τι να κάνουμε, να διακόψουμε για λίγο. <laughs> Συνάδελφοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε στη Συρία. Έχουμε καλέσει τον ε, κύριο Ιγκ Μιγκαρελή, τον οποίον ήδη έχω ε, αναφέρει, καθώς επίσης ε, και την αυτού εξοχότητα, τον κύριο Σελίμ Γενέτ, πρεσβευτή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξέρουμε πόσο δραματικά συνδέθηκε η χώρα αυτή, η Τουρκία, με την Συρία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το πρόβλημα των αμάχων είναι εξαιρετικά μεγάλο και διαρκώς διονγκούται ανεξάρτητη δημόσια ε, αρχή ερεύνηση στην ε, Συρία ε, απεσταλμένη και των, του Ηνωμένου, συγγνώμη, των Ηνωμένων Εθνών κατέδειξαν το εύρος της καταστροφής. Όλο και περισσότεροι είναι οι άμαχοι, άμαχοι οι οποίοι σκοτώνονται. Πάρα από 90.000 είναι αυτοί οι άμαχοι οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους και γίνονται πλέον καθημερινά επιδρομές κατά των πολιτών. Πλέον είναι πολλοί οι πολίτες, ε, οι πρόσφυγες οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια. Και πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει επιπλέον 50 ε, εκατομμύρια σε ανθρωπιστική βοήθεια για την προστασία των αμάχων στην ε, Συρία. Πρόκειται ένα ζήτημα ε, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα ε, με πολιτικό τρόπο. Χρειάζεται δημοκρατική μετάβαση όχι μονάχα για το καλό της ε, Συρίας και του Συριακού πληθυσμού, αλλά και για τη σταθερότητα στην περιοχή. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον κύριο Μιγκαρελή, Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τη Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Αραβική Χερσόνησο, Ιράν, Ιράκ και για να μας πει ποια είναι η δράση της εξωτερικής, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης να μιλάει ενώπιον της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για αυτή τη δραματική κατάσταση. Όπως ξέρετε, οι εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση έχουν διτό σκοπό πρώτον να, ε, να δώσουν ένα τέλο σε αυτές τις σφαγές γιατί είπατε ότι οι αριθμοί τρομάζουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερο από 25.000 νεκροί και ταυτοχρόνω βεβαίω πρέπει να βρεθεί η πολιτική λύση έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η σφαγή και έτσι ώστε να ανακουφιστούν όλοι αυτοί οι πληθυσμοί που υποφέρουν. Για να γίνει αυτό η ε, ε, και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίες Εξωτερικής Δράσης έχουν προσπαθήσει να ενεργήσουν βάσει εννέα αξώνων τους οποίους σύντομα θα αναφέρω. Πρώτον, να ανακουφιστούν οι πληθυσμοί. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Γνωρίζετε βεβαίως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα είναι ο πρώτος χορηγός ε, με ένα σύνολο 220 εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθυμίζω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ο πρώτος δωρητής γενικά ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά αυτό δεν αρκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εντείνει τις προσπάθειές της έτσι ώστε να βοηθήσει και τους εκτοπισμένους στο εσωτερικό της Συρίας αλλά ταυτόχρονα και τους πρόσφυγες που βρίσκονται σε τρεις ομόρες χώρες, η Ορδανία, Λίβανο και Ιράκ. Επί των δύο αυτών μετώπων λοιπόν θα υπάρξει ενισχυμένη προσπάθεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να είμαστε αποτελεσματικοί βεβαίως θα πρέπει να έχουμε καλύτερο συντονισμό της βοήθειας που δίνουν οι διάφοροι δωρητέ, και για να το κάνουμε αυτό την επόμενη εβδομάδα ενδεχομένως στη Νέα Υόρκη θα λάβει η χώρα συνάντηση, συνεδρίαση των, ε, των δωρητών υπό την Επίτροπο κυρία Γεωργίευα έτσι ώστε να αποφασιστεί αφενός η αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ε, κυρίως δεν να κινητοποιηθούν οι χώρες του κόλπου, οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν ε, σταθεί στο ύψος ε, των καταστάσεων και αφετέρου για να ενισχυθεί ο συντονισμός. Βεβαίως φτάνει και το ο χειμώνα και γνωρίζετε ότι οι εκτοπισμένοι και οι πρόσφυγε υποφέρουν περισσότερο το χειμώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για μα να δράσουμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα για να βοηθήσουμε αυτούς τους δυστυχείς. Δεύτερο άξονα είναι η στήριξη προ τι γειτονικέ χώρε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια γιατί γνωρίζετε ότι στην Ιορδανία, στην Τουρκία ήδη υπάρχουν στρατόπεδα. Στον Λίβανο και την Ιορδανία υπάρχουν πρόσφυγε που ζουν σε αστικέ περιοχέ και βεβαίω θα πρέπει να βοηθηθούν αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε κυρίως ε, ε, την Ιορδανία και το Λίβανο, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο πολιτική αποσταθεροποίησης. Η Ιορδανία και ο Λίβανος για λόγους που γνωρίζετε όλοι, είναι ευάλωτες, ευαίσθητες χώρες ε, και επομένως θα πρέπει να κάνουμε ό,τι γίνεται περισσότερο ότι είναι δυνατόν έτσι ώστε να μην υπάρξει πολιτική αποσταθεροποίηση. Αυτός είναι ένας προσφυλής στόχος, τον οποίο θα επιδιώξουμε τον, τους τις επόμενες ημέρες έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές ε, και έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, στις χώρες τις οποίες ανέφερα προηγουμένως να δώσουμε ε, βοήθεια όσον αφορά ιατροφαρμακευτικό υλικό αλλά και όσον αφορά και την εκπαίδευση. Στην Βηρητό θα πρέπει να δώσουμε όλες τις, καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες έτσι ώστε να μην υπάρξει πολιτική αποσταθεροποίηση λόγω της μαζικής ροής προσφύγων. <clears throat> Τρίτη προσέγγιση. Είναι η στήριξη ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών αυτή τη στιγμή και τα Ηνωμένα Έθνη και ε, ο Αραβικός Σύνδεσμος προσπαθούν να συνεργαστούν. Ε, εμείς ε, στηρίζουμε τον Κόφι Ανάν και η στήριξη αυτή βεβαίως είναι στη διάθεση και του Κάρι Μπραχίμη. Επανειλημμένα έχουμε μιλήσει μαζί τους. Η Πατή εκπρόσωπος και την επόμενη εβδομάδα στην ε, Νέα Υόρκη θα συναντήσει και τον πρόεδρο Αλαράμπη και έχουμε πει επανειλημμένα, έχουμε πει επανειλημμένα ότι εμείς θέλουμε παρουσία των Ηνωμένων Εθνών στη Δαμασκό και γνωρίζετε ότι και εμείς αλλά και τρεις πρεσβείες ε, των ε, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι στη διάθεση του Αχτάρ Μπραχήμι έτσι ώστε να του παραχθεί όλη η απαραίτητη βοήθεια τέταρτος άξονας της παρέμβασής μας. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, αυτή η αντιπαράθεση χρονίζει είναι η διάσπαση της αντιπολίτευσης. Η ύπατη εκπρόσωπος, καθώς επίσης και όλες οι υπηρεσίες, ευρωπαϊκές υπηρεσίες εξωτερικής δράσης, έχουν αναλάβει δράση έτσι ώστε να πείσουν την αντιπολίτευση να δημιουργήσει μια κοινή πλατφόρμα, να προετοιμάσει δηλαδή την μετά Άσαντ εποχή. Βεβαίως εμείς δεν τους ζητούμε να ενωθούν γιατί αυτό θα ήταν παράλογο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικές ιδεολογίες, οποίες έχουν διαφορετικά δόγματα και φυσικά έχουν κάθε δικαίωμα να παραμείνουν στις πολιτικές θέσεις που θέλουν. Αλλά βεβαίως αν θέλουν να προετοιμάσουν την μετάβαση θα πρέπει να το κάνουν μέσω της προετοιμασίας μιας κοινή πλατφόρμας. Οργανώσαμε λοιπόν επανειλημμένα πολλές συναντήσεις με τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, κυρίως δε και πρωτίστως με το Συριακό Συμβούλιο, έτσι ώστε, Εθνικό Συμβούλιο, έτσι ώστε ε, να ε, θέσουμε στη διάθεσή τους την τεχνογνωσία που έχουμε και βεβαίω στηρίζουμε πλήρως ε, και τον Ελλαδικό Σύνδεσμο, ο οποίο επανειλημμένα ε, ε, συνένωσε και συνεδρίασε στο Κάιρο με όλους τους εκπροσώπους. Βεβαίω θέλουμε να καθησυχάσουμε και όλες τις μειονότητε. Είναι γεγονός ότι όλες οι μειονότητε, κυρίως οι, οι, οι Αλαουιστές και οι Χριστιανοί, φοβούνται την ε, μετα-Άσαντ εποχή, φοβούνται δηλαδή ότι θα υπάρξει ε, ένα κυνήγι μαγισσών ε, μετά το τέλος της περίοδου Άσαντ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμε να υπάρξει σωστή αντιμετώπιση όλων των μειονοτήτων. Ο επόμενος άκρος της δράσεις μας είναι να καλύψουμε τις πηγές τροφοδοσίας της κυβέρνησης. Πριν από μια εβδομάδα περίπου συναντήθηκαν οι Υπουργοί Εξωτερικών στην Κύπρο και μας ζήτησαν ε, να αναλάβουμε, να πάρουμε μια σειρά επιπλέον ε, κυρώσεων, επιπλέον δηλαδή αυτών που έχουμε ήδη πάρει, έτσι ώστε να μην ε, υπάρξει πλέον τροφοδοσία της, του καθεστώτος Ασάντα και έτσι ώστε αυτή η μηχανή θανάτου να σταματήσει να λειτουργεί. Αυτό το μεταφέρουμε σε όλους τους εταίρους μας. Γνωρίζετε ότι μια σειρά φόρα έχουν ε, διοργανωθεί έτσι ώστε να προετοιμαστεί η πολιτική μετάβαση. Πρώτον, οι φίλοι της Συρίας με μια σειρά συναντήσεων και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα και στο Παρίσι. Θα υπάρξει σίγουρα και την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ε, μια συνάντηση της πυρηνικής ομάδας Core Group των φίλων της Συρίας υπό την Προεδρία της Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων ΗΠΑ. Ε, επίσης ε, υπήρχε αυτή η συνάντηση που έγινε μία φορά στη Γενέβη και η οποία αφορούσε χώρες ε, οι οποίες είναι δύσκολο να τις αγγίξουμε εμείς όπως ας πούμε η Ρωσία. Αλλά πρέπει να διατηρηθεί και αυτή, αυτός ο δίευλος επικοινωνίας ανοιχτός και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία του Αιγυπτίου Προέδρου που αποφάσισε να συνενώσει τους Σαουδάραβες τους ε, Τούρκους, τους Ιρανούς, ένα κουαρτέτο δηλαδή το οποίο θα μπορούσε ε, να ε, πείσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τον Άσαντ ότι πλέον τελείωσε η δικιά του, το δικό του καθεστώς και ότι θα πρέπει να περάσει την εξουσία στους, στην αντιπολίτευση. Γνωρίζουμε ότι η Σαουδέλ Φεϊζάλ ε, δεν ε, είναι καλά στην υγεία του, αλλά ενδεχομένως ε, δεν είναι μόνο πρόβλημα της υγείας του πρίγκιπος ο λόγος για τον οποίο η Σαουδική Αραβία δεν συμμετείχε σε αυτήν την συνεδρίαση. Ξέρετε πάντως ότι η Αίγυπτος, το Ιράν, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία είναι αυτοί οι τέσσερις πρωταγωνιστές οι οποίοι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, μπορούν να είναι οι μοχλοί οι οποίοι θα κινήσουν ενισχύσουν την ε, διαδικασία. Και επομένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρωτοβουλίε των χωρών αυτών και βεβαίω ε, θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι μπορούν να συζητήσουν μεταξύ του. Υπάρχει και ένα έβδομο άξονας ο οποίος μας έχει ζητηθεί από πολλές χώρες μέλη και θέλουμε να τον ε, ακολουθήσουμε είναι ο άξονας ο οποίος σχετίζεται με την λογοδοσία και με την ευθύνη ε, όσων έχουν ε, κάνει ε, πράξεις εγκληματικές. Είπαμε ότι δεν θα υπάρξει ατιμορρησία. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρξει προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ξέρετε ότι εδώ δεν πρέπει να το κρύψουμε. Είναι... Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό ενδεχομένως εάν ε, επικράμεται επί της κεφαλής του Ασάντ ε, το ποινικό δικαστήριο της Χάγης, ίσως λέω να μην είναι ο καλύτερος τρόπος για να τον πείσει κανείς να φύγει, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό και αυτό που είναι βέβαιο και από αυτού ήταν πάρα πολύ σαφής και η εκπρόσωπος ε, είναι ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε ατιμορρησία για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και η Διεθνής Επιτροπή η οποία έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της, ε, των Ηνωμένων Εθνών στη Γενέβη ε, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ε, τα, ε, ότι είναι απολύτως σαφές ή τουλάχιστον υπάρχουν σαφέστατες ενδείξεις ότι στην ε, Συρία το καθεστώς έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Είναι γεγονός πάντως επίσης ότι και στην αντιπολίτευση υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αίμα στα χέρια τους. Δεν έχουν, δεν έχουν συμπεριφερθεί και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, έλεγα και προηγουμένως ότι δουλεύουμε με τους φίλους της Συρίας. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν μαζί με τους φίλους της Συρίας ε, μία ομάδα η οποία ασχολείται με την ανασυγκρότηση της Συρίας ε, σε συνεργασία και με την Γερμανία. Συμμετέχουμε και εμείς σαν Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Στόχος των, της ομάδας αυτής είναι η εκτίμηση, η αξιολόγηση των ζημιών που έχουν γίνει στην Συρία και επομένω να γίνουν κάποιοι υπολογισμοί όσον αφορά την ανασυγκρότηση τη χώρα αυτή, έτσι ώστε να μην βρεθούμε προεκπλήξεων την επόμενη μέρα. Και ο ένατος άξονας, και εκεί θα σταματήσω, είναι βεβαίως το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μεγάλο άγχος υπάρχει ε, στα Ηνωμένα Έθνη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων ε, Εθνών δεν ήταν σε θέση να καταλήξει σε κάποιο ψήφισμα. Γνωρίζουμε όλοι τους λόγους ε, και επομένως θα ήθελε να υπάρξει ένα ψήφισμα το οποίο θα καταδικάζει τις πρακτικές του Άσαντ ε, και τις εγκληματικές του ενέργειες. Ε, γνωρίζετε ότι σε επίπεδο διεθνούς δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν δύο χώρες οι οποίες είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, και που συνεπικουρούμενοι και από τα BRICS που δεν είναι από τις χώρες BRICS που δεν είναι και πολύ ζεστές για ένα τέτοιο ψήφισμα δεν, δεν καταλήγουν. Βεβαίως γίνεται προσπάθεια συνεργασίας του Σεργέ Λαυρόφ και με την Κίνα έτσι ώστε να σφυριλατηθεί μια τέτοια κατάσταση στο, στο, στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, έτσι ώστε να υπάρξει ένα ψήφισμα καταδικαστικό. Αυτά ε, είναι, αυτοί είναι οι, έξι, η συγγνώμη, οι εννέα άξονες επί των οποίων εργάζεται, είπατε, εκπρόσωπος ε, με την Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης. Υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν προσκόμματα. Γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Θα δούμε πώς θα έχει η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Μπράβο σας, όπως πάντα, εξαιρετικός. We κύριε Πρέσβη, θέλουμε τη βοήθειά σας για τη συζήτηση του θέματος των σύρων προσφύγων στα σύνορα με τη Συρία και τι αντίκτυπο ε, έχει ε, στην Τουρκία, στη χώρα σας, η έλευση των προσφύγων. Ποιες είναι οι απόψεις της τουρκικής κυβέρνησης για το πώς θα τερματιστούν οι σφαγές στη Συρία και να επέλθει ένας ε, γνήσιος δημοκρατικός μετάβαση, μάλλον, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω ενώπιον των αξιότιμων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω τον προελίσαντα, αλλά να απηχήσω στη δική μου ομιλία κάποια τμήματα της παρέμβασής του και να σε εξηγήσω πώς εκλαμβάνουμε εμείς την κατάσταση στην Ταρκία. Έχουμε διδυτή ανησυχία, μία για τη Συρία και γενικότερα για την ευρύτερη περιοχή και ε, ανησυχία επίσης για την ίδια την Τουρκία. Δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση μάλλον θα επιδεινωθεί. Ε, βλέπουμε ε, δολοφονίες, ε, βιοπραγίες καθημερινά και είμαστε σε απόγνωση. Το καθεστώς κάνει απονενοημένα πράγματα και είναι, δεν είναι προβλέψιμο εκ τούτου και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στις μελλοντικέ μας δράσεις. Μας ανησυχεί η επόμενη μέρα τι θα συμβεί όταν τελειώσουν όλα αυτά. Είδαμε σε άλλε χώρε τη περιοχή ε, τι έχει συμβεί και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα. Ε, παραδείγματος χάρη να υπάρξουν διαχωρισμοί στο εσωτερικό της ε, κοινωνίας ε, της Συρίας λόγω των θρησκευμάτων παραδείγματος χάρη έχουμε μεγάλο αριθμό προσφύγων ε, στην ε, Τουρκία και το σημαντικότερο για μας ε, είναι το ζήτημα της εδαφικής ακαιρεότητας. Χρειαζόμαστε επίσης ένα μεταβατικό σχέδιο για την μετά Ασάντ εποχή. Θα ήθελα να επαναλάβω μόνο το ότι δεν θέλουμε λόγω εθνοτικής προέλευσης ή θρησκευτικών διαφορών να διχαστεί η κοινωνία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να στηρίξουμε την αντιπολίτευση. Αλλά όλοι ξέρουν ότι δεν υπήρχε ποτέ αντιπολίτευση και είναι πολύ δύσκολο να οργανωθεί μια αντιπολίτευση. Πολλοί μένουν στην αλλοδαπή. Όσοι ε, αγωνίζονται στο εσωτερικό της χώρας δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με όσους είναι στην αλλοδαπή. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να ενωθούν και να μην αποκλείσουμε κανέναν. Η αντιπολίτευση θα πρέπει να συναπαρτίζεται από όλες τις ε, ομάδες ομάδες, ε, ε, πολιτικές, θρησκευτικέ και κοινωνικές ε, της χώρας. Έχουμε ήδη καταβάλει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, ελπίζουμε να καρποφορήσουν σε σχέση τώρα με την διεθνή κοινότητα. Όλοι ε, καταγγέλουν αυτά τα ομά εγκλήματα, αλλά είναι δεμένα τα χέρια μας και δεν μπορούμε να κινηθούμε. Ε, Τά εδώ και πάρα πολύ καιρό όχι μόνο τις ε, κυρώσεις ε, αλλά και συγκεκριμένη δράση για να προστατεύσουμε ε, η μη τι άλλο τους εσωτερικά εκτοπισμένους Σύρους. Υπάρχουν κάποιες χώρες που αντιτάσσονται σε τέτοιου είδους δράση και ελπίζουμε ότι τελικά θα συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να είναι στο σωστό στρατόπεδο της ιστορίας. Ε, στην Τουρκία, όπως σας είπα, υπάρχουν πάνω από 80.000 ε, εσωτερικά εκτοπιστέντες ε, και είχαμε φτάσει στις 120.000, αλλά περίπου 38.000 επέστρεψαν. Έχουμε 12 περίπου στρατόπεδα, 8 υπάρχουν και 4 οικοδομούνται τώρα. 60.000 ανθρώπους ε, υποδεχόμαστε και περιμένουμε να οικοδομήσουμε και άλλα στρατόπεδα για να υποδεχτούμε και άλλες 40.000. Δεν ξέρουμε για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν εκεί. Πλησιάζει και ο χειμώνα και μπορεί κάποιοι να σκέφτονται «Α, τι χώρα είναι ε, η Τουρκία, αλλά είναι δρυμής ο χειμώνα ε, και πραγματικά μπορούν να κατέβουν πολύ οι θερμοκρασίες το χειμώνα. Πρέπει να προετοιμαστούμε για όλη τη διαμονή, όποια και αν είναι αυτή, των προσφύγων και να προσφέρουμε υπηρεσίες όλων των ειδών, ε, κοινωνικές υπηρεσίες, ε, ε, ιατρικές υπηρεσίες, ακόμη και το πρόσβαση στο διαδίκτυο. 12 εκατομμύρια έχουμε ήδη δαπανίσει για τους πρόσφυγες. Επίσης υπάρχουν συγγενείς ε, πέρα από τη Μεθόριο και δεν είναι όλοι μέσα σε στρατόπεδα, αλλά ε, υπάρχουν και σε κάποιες τουρκικέ πόλεις και φυσικά είναι ε, ευπρόσδεκτοι η αρρωγή της διεθνούς κοινότητας ε, δεν επαρκεί. Πρέπει να το πούμε. Ξέρουμε ότι όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε γειτονικέ χώρες όλοι έχουν συνεισφέρει αλλά μπορεί να κάνει περισσότερα ε, η διεθνής κοινότητα. Είμαστε σε επαφή με την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες ε, του ΟΗΕ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια σχέδια από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευπρόσδεκτη είναι οποιαδήποτε βοήθεια ε, ακόμη και μέσω της ΕΚΟ. Ε, ε, αυτή τη στιγμή η βοήθεια από μεμονωμένες χώρες δωρητές είναι αυτό που χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια, μπορέσαμε να διαχειριστούμε την κρίση, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για τα χειρότερα. Μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο η κατάσταση, μπορεί να έρθουν και άλλοι πρόσφυγες. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τους σύρους που βρίσκονται σε μεθοριακές περιοχές ε, προτού βγουν από τη χώρα, να τους ε, ε, προσφέρουμε τα απαιτούμενα τρόφιμα και άλλα είδη καθημερινά που χρειάζονται στα σύνορα της ε, Τουρκίας ε, με τη Συρία προτού τα διασχίσουν. Ε, ένα άλλο θέμα είναι η τρομοκρατία στη χώρα μας, το οποίο και περιθάλπτεται, υποθάλπτεται συγγνώμη, και υποβοηθείται από την κυβέρνηση και ε, μιλώ φυσικά για τη Συριακή κυβέρνηση και χρησιμοποιούν ε, ε, το PKK εναντίον μας. Δημιουργείται θέμα ασφαλείας πλέον για την Τουρκία και πιστεύω ότι ε, για να μπορέσουμε να δράσουμε ουσιαστικότερα χρειαζόμαστε τη διεθνή κοινότητα. Ε, οδήποτε δράση πρέπει να έχει εγκριθεί από το ΝΟΙΕ. Ο δάλος ε, δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί. Όπως είπε και ο κύριος Μιγκαρέλη, ε, είναι δυνότατη η κατάσταση. Είναι... ντροπή και έσχος ε, ε, ε, να βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα. Θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Κατά βάση πιθανότητα θα τα καταφέρει από μόνη η αντιπολίτευση, αλλά πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε. Ομά εγκλήματα διεπράχθησαν παντού. Έχουμε όλο ένα και λιγότερε πληροφορίε για το προξενείο και οι πρεσβεία μα έχουν κλείσει στη Συρία. Από τον τύπο ότι μαθαίνουμε ουσιαστικά και δεν πρόκειται, ξαναλέω, να βελτιωθεί η κατάσταση. Μπορεί κάποιο να πει ότι δεν είναι η ίδια η κατάσταση όπως ε, στη Βόρεια Αφρική. Μάλλον θα διαρκέσει περισσότερο το πρόβλημα στη Συρία και θα δημιουργήσει μεγαλύτερε έγνοιε, ανησυχίες και προβλήματα για σας, για μας. Ε, πρέπει να σπεύσουμε, να δράσουμε, να σταματήσω καλύτερα και να απαντήσω και σε ερωτήσει αν υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Έχω έναν ε, κατάλογο τεσσάρων αγορητών που έχουν ζητήσει να παρέμβουν. Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Α, πέντε. Πέντε είναι οι ομιλητές. Έξι, ενάμιση λεπτό, κατεβαίνει ο μέσος Και εγώ θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Μία ερώτηση στον δόκτωρα Μιγκαρέλη. Δόκτωρα Μιγκαρέλη, μιλήσατε για κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης. Τα όρια όμως των ομάδων της αντιπολίτευσης είναι ασαφή. Ερώτηση λοιπόν έχετε σφυγομετρήσει την πραγματική βούληση συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ομάδων και αν ναι υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, συγκεκριμένοι στους οποίους θέλουν να συνεργαστούν. Γιατί είδαμε τι έγινε στην ε, Λιβύη. Διώξανε τον Καντάφη και μετά... Ε, βρήκαμε μπροστά μας μία σειρά γκρουπούσκουλα τα οποία ήθελαν να γίνουν ας πούμε οι αφέντες της περιοχής. Επομένως να μην διατρέξουμε τον ίδιο κίνδυνο. Προς τον πρέσβη της Τουρκίας να ρωτήσω το εξής. Φαντάζομαι ότι θα σας έχει περάσει από το μυαλό και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Ποια νομίζετε ότι θα ήταν η διάθεση των αραβικών χωρών να παρέμβουν έτσι ώστε να δημιουργηθεί απαγόρευση υπερπτήσεων στη Συρία, δηλαδή no-fly zone. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκόμες. 1,5 λεπτό. Εγώ δεν ξεπέρασα το 1,5 λεπτό, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μεγκαρέλη για την ε, τοποθέτησή σα. Πολύ καλή. Θα ήθελα να σα ρωτήσω τώρα. Εμείς Πώς θα υποστηρίξουμε τον κύριο Μπραχήμι, όχι μόνο με την επιμελητία ε, πολιτικά, πώς θα είμαστε ένα τμήμα της ομάδας του στα διαβήματα που κάνει. Ε, το έχετε σκεφτεί αυτή. Δεύτερον, το Ιράν είναι πρωταγωνιστής, υποστηρίζει τον Ασάντ, κάνουμε εμείς τίποτα με το Ιράν. Εντάξει για τα πυρηνικά, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το Ιράν και να τους θέσουμε και το θέμα του Ασάτ. Δεν θα ήταν ε, ε, σκόπιμο και χρήσιμο κάνουμε τίποτα προς τα εκεί. Στη συνέχεια, διερευνούμε ε, τη δυνατότητα να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας στον ΟΗΕ, διότι η τραγωδία στη Συρία ποια είναι. Το είπε μόλις και ο πρέσβης της Τουρκίας. Τώρα είναι η Συρία, αύριο μπορεί να είναι πολλά άλλα μέρη. Αν δεν σταματήσει το βέτο και το μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και βεβαίως η Κίνα και η Ρωσία παίζουν πολύ αρνητικό ρόλο, ιδιαίτερα η Ρωσία. Αλλά τι γίνεται με τη Βραζιλία και την Ινδία. Δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί τους για τις μεταρρυθμίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τη διεύρυνσή τους. Μπορεί να αλλάξει η κατάσταση ε, γίνει κάτι τέτοιο. Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή για τη στρατιωτική ε, ε, ε, εκδοχή. Αν η χώρα σας απειληθεί ακόμα περισσότερο από όσο απειλείται σήμερα. Χρειάζονται αντιαεροπορικά τώρα. Αυτό χρειάζεται. Γιατί ο, ο Ασάντ επιτίθεται τώρα από αέρος. Και αυτό θα έχει και επιπτώσεις εκτός του ΠΚΚ, μήπως όλα αυτά σφυριλατήσουν την ενότητα του σύνολου κουρδικού ε, έθνους. Ρωμέβα Λόπες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Μιγκαρέλη και να τον ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ε, ότι καταβάλλεται με αλφαγιώτα κάθε δυνατή προσπάθεια για να ε, αποτραπεί η σφαγή η Σύμβαση της Γενέβης εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους, αλλά και τους εχμαλώτους πολέμου και την άμαχο πληθυσμό. Υπάρχουν συμβάσεις της Γενέβης που έχουν υπογράψει πάρα πολλές χώρες. Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, πού βρίσκεται ακριβώς. Ο κόσμος έχει τρομακρατηθεί ε, από ό,τι συμβαίνει. Αλλά είναι βαρβαρότητα αυτά. Είναι εποχές πριν τη σύμβαση της Γενέβης. Ε, τώρα γιατί δεν υπάρχει ένα ψήφισμα για να γίνεται σεβαστό το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Γιατί δεν μπορούν οι χώρες αυτές να διαφωνήσουν με ψήφισμα το ΟΗΕ για την εφαρμογή και το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε εκεί για να σταματήσουν οι σφαγές που είναι το πρώτο. Αυτό προτεύει, να σταματήσει ε, η σφαγή του αμάχου πληθυσμού. Δεν θα μπορούσαμε να επιμείνουμε εκεί για να είναι πιο αποτελεσματική η δράση μας. Τι γίνεται όταν δεν σέβονται χώρες στη Σύμβαση Γενέβης, υπάρχουν ψηφίσματα, τι προβλέπουν τα Ηνωμένα Έθνη. Με την πρόφαση ότι εντάξει κάνει ε, βιαιότητες και ε, ομότητε και η αντιπολίτευση, αυτό δεν είναι επιχείρημα, αυτό είναι φιλοσοφία του πολέμου. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Miss Lösing. Η κυρία Ja, vielen Dank. Ich stimme mit meiner... Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την προλαλή Η σφαγή θα πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει, να αποτραπεί. Ε, ε, είναι απολύτως απαραίτητο. Και βεβαίως κάθε σφαγή είναι καταδικαστέα. Δεν συμφωνώ όμως με την παρατήρηση ότι δεν είναι επιχείρημα ε, ή ότι δεν είναι σημαντικό ότι τα ίδια κάνει και αντιπολίτευση και ε, παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και σφαγιάζει επίσης. Πολλοί συνάδελφοι ε, τα παρουσιάζουν διαφοροποιημένα, ότι υπάρχουν, ξέρετε, διάφορες ομάδες της αντιπολίτευσης. Παρόλα αυτά, απέναντι ε, είναι το καθεστώς και γίνεται πάντα λόγος για το καθεστώς και την αντιπολίτευση. Μπλοκ. δεν υπάρχει δυνατότητα πλέον λύσης μέσα από διαπραγμάτευση ή από συζήτηση, αλλά παρόλα αυτά θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει δυνατότητα ειρηνικής επίλυσης με διαπραγματεύσεις. Έχει εξαφανιστεί αυτή. Στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, τη γερμανική, χτε δημοσιεύτηκε ένα άρθρο που έλεγε ότι η ύπατη αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα απευθύνθηκε και ε, στη ε, Συριακή κυβέρνηση και στους εξεγερθέντες και τους έχει ε, ε, συλλητεύσει για μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η κυβέρνηση στρατολογεί παιδιά, ας πούμε, και οι εξεγερθέντες επίσης κάνουν πολλές βιοπραγίες, δεν χρειάζεται να επεκταθώ εδώ, αλλά υπάρχει καμιά λύση. Προς τα πού στρεφόμαστε, ακόμα και τη στρατιωτική επέμβαση. Και θα ήθελα να σας αποτρέψω από αυτό. Δεν μπορούμε να είμαστε υπέρ μιας τέτοια επέμβαση. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, πώς θα γίνει. Σήμερα το πρωί είχαμε συνομιλίες με εκπροσώπους της Σαουδική Αραβίας που μας είπαν ξεκάθαρα ότι υποστηρίζουν Ισλαμιστικέ δυνάμεις και μπορούμε να φανταστούμε και σε ποια κατεύθυνση θα πάνε ε, αυτά και πού θα στραφεί η χώρα. Λοιπόν, ερωτώ και πιεστικά ποια είναι η δημοκρατική προοπτική στην οποία εμείς προσβλέπουμε και ποιο ενδεχόμενο διενήγεται, τι δυνατότητες βλέπουμε. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. One minute and a half. Ενάμιση λεπτό. Ε, θα ήθελα και εγώ καταρχήν να καταγγείλω με τον πιο έντονο τρόπο τις σφαγές που λαμβάνουν χώρα στην Συρία ιδιαίτερα σφαγές αμάχων και παιδιών, γυναικοπαίδων. Δεν μπορεί αυτό παρά να σπρώχνει κάποιον να σκέφτεται ότι πρέπει να υπάρξει μια λύση. Καταλαβαίνω βέβαια ότι η σύγκρουση που υπάρχει είναι τόσο σφοδρή μεταξύ αντιπολίτευσης ή δυνάμεων της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης που δυσκολεύει κάποιον να καταλήξει σε, ένα σε μια συγκεκριμένη απόφαση για το τι πρέπει να κάνει. Έχω όμω μια ερώτηση και στον κύριο Μικαρέλη και στον πρέσβη τη Τουρκία, γιατί βρίσκω μια μεγάλη αντίφαση στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα. Στη Συρία υπάρχει η αντίδραση, όπω την ξέρουμε, τη αντιπολίτευση και υπάρχει η σφοδρή βαρβαρότητα εκ μέρου του κράτου για να καταστήλει ε, αυτή την ε, εξέγερση. Στην Τουρκία υπάρχει κάτι ανάλογο. Μια μερίδα του πληθυσμού αντιδρά, μιλώ για τους αντάρτες του ΠΚΚ και το κράτος αντιδρά κατά τον τρόπο που αντιδρά ε, το κράτος της Συρίας. Πώς γίνεται αυτή η αντίφαση. Στη μια περίπτωση είναι αντιπολίτευση εξεγερμένη, αναζητά τα δημοκρατικά της δικαιώματα. Δεν είναι το ίδιο που συμβαίνει και στην Τουρκία. Γιατί στη μια περίπτωση παίρνουμε τη θέση υπέρ, του, ε, υπέρ της αντιπολίτευσης και στην άλλη περίπτωση υπέρ του κράτους. E Ευχαριστώ κύριο Λίζεκ από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε για το μέλλον. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τον κύριο Μιγκαρέλη, όμως η κατάσταση πώς έχει ε, σήμερα ως εξής. Πρέπει να σταματήσουμε αμελητή τη σφαγή. Έχει κλιμακωθεί η σύραξη ανάμεσα στο καθεστώς Ασάντ και την αντιπολίτευση σε βαθμό που φαίνεται ότι μόνο με στρατιωτικά μέσα μπορεί να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτή την κατάσταση και ρωτώ γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι, πόσα πολεμοφόδια, πόσα μέσα έχει ο πρόεδρος Ασάντ, έχει στρατιωτική υποστήριξη, τροφοδοτείται ο στρατός του ε, σε πολεμοφόδια ή λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη βοήθεια και από ποιον έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Θα ήθελα να ρωτήσω τον πρέσβη το εξής. Ποια είναι η κατάσταση για τους ε, σωματικούς ε, ελέγχους ε, που γίνονται στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία. Ποιος ελέγχει ακριβώς τα σύνορα στη πλευρά της Συρίας. Ελέγχεται το κομμάτι αυτό από την κυβέρνηση ή από τους αντάρτες, από την αντιπολίτευση. Ευχαριστούμε κυρία Λαβέλα. Τζαβέλα. Ευχαριστώ τους ομιλητές για την συνεισφορά τους στη συζήτηση. Η ερώτησή μου προς τον κύριο Μέγκελ είναι έχει αξιολογηθεί η ευρωπαϊκή μας παρέμβαση στη Βόρειο Αφρική. Από ό,τι βλέπουμε τώρα, μετά την Αραβική Άνοιξη έχουμε το Αραβικό Φθινόπορο. Υπάρχει μία εξέγερση σε όλο το μουσουλμανικό κόσμο στο Νότο, άρα κάτι δεν πήγε καλά. Θέλουμε να δούμε τη Συρία σε κατάσταση, στην κατάσταση που είναι και η Λιβύη αυτή τη στιγμή 500 ε, ένοπλες ομάδες γυρίζουν στη Λιβύη λαιλατώντας, βιάζοντας και κάνοντας οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Είναι αυτό ένα κράτος δικαίου το οποίο στεριώσαμε. Κύριε Πρέσβη, είστε κοντά, ξέρετε τι γίνεται. Ποιοι είναι αυτοί που προμηθεύουν και τις δύο πλευρές για να έχουμε ένα εμφύλιο στη Συρία. Είναι εμφύλια σύραξη. Μπορούμε να διακινδυνεύσουμε πάλι μια διεθνή παρέμβαση. Αυτό εννοείται ότι είναι τα χέρια μας δεμένα, πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Τι παραπάνω, διεθνή παρέμβαση και μετά τον Άσαντ τι, σαν την κυβέρνηση που βάλαμε στη Λιβύη, σαν αυτά που βλέπουμε να γίνονται τώρα στην Τινησία. Μόνο η Αίγυπτος προσπαθεί να βρει το βηματισμό της. Έχουμε κάποια, κάποια συγκεκριμένη αξιολόγηση της ευρωπαϊκής μας πολιτικής μετά από όλα αυτά που είδαμε να γίνονται. Ευχαριστώ κύριε Φραντσίσκα Μπράντνερ. Ευχαριστώ πρέπει να πω ευθύ εξ αρχή ότι δεν ήμουν από την αρχή τη παρουσίασή σα. Είχαμε ε, κάποιου εκπροσώπου, αξιωματούχου από τη Λιβύη ε, και ζητώ συγγνώμη αν ρωτήσω κάτι το οποίο έχετε ήδη απαντήσει. Για ε, τους πρόσφυγες. Ακούμε πολλές φήμες ότι η ε, βοήθεια που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ερυθρού Σταυρού δεν φτάνει εκεί που πρέπει, αλλά φτάνει σε λάθος χέρια, ε, σε αντάρτες ενδεχομένω που εξοπλίζονται, αλλά όχι ως ανθρωπιστική βοήθεια. Όπως ε, ε, είπα, είναι φήμες, αλλά μήπως ο ρόλος της Ερυθράς Μισελίνου εκεί είναι προβληματικός, γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα επιτόπου. Η πρώτη ερώτηση. Και ένα δεύτερο τα δεδομένα στην περιφέρεια, δεν ξέρω πώς το είπατε στα αγγλικά, ε, θα άλλαζαν πάρα πολύ αν άνοιγε το Ισραήλ τα σύνορά του για πρόσφυγες. Εμείς μήπως θα πρέπει να το ζητήσουμε κάτι τέτοιο, να πιέσουμε ή να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ αυτού, γιατί μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, γίνεται αντιληπτή η χώρα στην περιοχή και το θεωρείτε σκόπιμο κάτι τέτοιο θετικό. Αυτές τις δύο ερωτήσει είχα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σαλαφράγκα. Τελευταίος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση την περασμένη εβδομάδα ε, στην Ολομέλεια με την ύπατη εκπρόσωπο, ε, όπου ακούστηκε όλη η απογοήτευση και όλη η ματέωση την οποία μας προκαλεί η κατάσταση. Ε, το ακούσαμε από συναδέλφους πάρα πολύ εύγλωτα στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι η κατάσταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας και το πρόβλημα που ζει η Ευρωπαϊκή Ένωση που αναλώνεται στα εσωτερικά της με την κρίση εμπιστοσύνης κτλ ο εκλογικός ορίζοντας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά μαζί λοιπόν κατά κάποιο τρόπο ε, δίνουν μια κατάσταση ευρεωμένη, πώς να το πω, ε, κάτι που δεν μπορεί να λυθεί με διεθνή παρέμβαση. Προσπαθεί ε, το καθεστώς να ε, πατάξει την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση βλέπει ότι δεν μπορεί να βοηθηθεί από τη διεθνή κοινότητα. Υπάρχει κρίση και στο Ιράν, ε, αλλά οι νεκροί πολλαπλασιάζονται και είναι πολλά τα χρήματα που δίνουμε για ανθρωπιστική βοήθεια και εγώ είπα στην ύπατη εκπρόσωπο ότι εμεί δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στο ρόλο του Διεθνούς Σταυρού, αλλά να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Και ρωτώ τον κύριο Μιγκαρέλη, υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουμε ανθρωπιστικό διάδρομο, όπως ζήτησαν κάποια κράτη-μέλη, να προσπαθήσουμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα απαγόρευσης ε, πτήσης. Ε, ακούσαμε τον Πάπα ε, στην επίσκεψή του στο Λίβανο να λέει τι συνέπειες έχει εξοπλισμός και των δύο πλευρών. Και τέλος θα πρέπει να υποστηρίξουμε σαφώς την ε, ε Τουρκία στην ε, ε, καταπολέμηση του ΠΚΚ και των ενόπλων ομάδων που κυκλοφορούν και στα σύνορα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνη της την Τουρκία να επομίζεται όλα τα αρνητικά αυτής της κρίσης και αυτής της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μιγκαρελή, παρακαλώ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε 7, 8 λεπτά. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους βουλευτές που έθεσαν ερωτήματα. Θα απαντήσω στα πιο σημαντικά ε, θέματα γιατί ε, πέρα από την συμμετοχή σε οποιαδήποτε ομάδα και τις επαφές που μπορούμε να έχουμε βεβαίως υπάρχουν και ζητήματα ε, πολιτικής τάξης τα οποία δεν είναι απλά. Όσον αφορά κύριε Πρόεδρε την ε, θέληση των ε, διαφόρων ομάδων της αντιπολίτευσης να συνεργαστούν. Υπάρχει κατακαιρματισμός ε, υπό πολλές έννοιες. Δηλαδή υπάρχει εσωτερική και εξωτερική αντιπολίτευση που δεν έχουν πάντα τις ίδιες θέσεις. Μια δεύτερη διαχωριστική γραμμή είναι αυτοί που θέλουν τον ένοπλο αγώνα, που θεωρούν δηλαδή ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο διαφραγμάτευσης με το καθεστώς αυτό και αντιθέτως αυτοί οι οποίοι ε, πιστεύουν ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα διαπραγμάτευσης και περαιτέρω πίεσης. Αυτή είναι μια σημαντική διαχωριστική γραμμή. Και υπάρχει και μια τρίτη διαχωριστική γραμμή που είναι βεβαίως ε, η θρησκευτική. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε θέση ε, αυτή η κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση να έχει κοινή πλατφόρμα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασίας, υπάρχει δυνατότητα να καταγραφούν τα κύρια πολιτικά χαρακτηριστικά της μετά Ασάτ περίοδου. Βεβαίως ε, θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς στις επαφές που έχουμε με την αντιπολίτευση. Αυτό προσπαθεί να κάνει και η Τουρκία στις επαφές που έχει με την αντιπολίτευση. Κάποια κράτη-μέλη που δουλεύουν με τον ίδιο σκοπό και βεβαίως ε, η ύπατη εκπρόσωπος γνωρίζεται ότι έχει ήδη οργανώσει συναντήσεις με ομάδες της αντιπολίτευσης βεβαίως. Δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να έχουμε κοινή πλατφόρμα. Όμως πέρα από τις διαχωριστικές γραμμές οι οποίες όντως υπάρχουν πιστεύω ότι μπορεί αύριο να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια κοινή πλατφόρμα δεν είναι απάντηση βασισμένη σε γεγονότα και συγκεκριμένα στοιχεία, είναι μια εκτίμηση. Δεύτερον, η ερώτηση της κυρίας ε, ε, ε ο ρόλος της Αλκάιντα, τι να σας πω, εγώ δεν έχω καμία πληροφορία από αυτού και επί τη βάση των εκθέσεων που διαβάζω αναφέρεται μερικές φορές ότι ε, ε, ε, κύτταρα της Αλκάιντα που ήταν παλιότερα σε γειτονικέ χώρες έχουν πλέον βάση στη Συρία αλλά δεν έχω την δυνατότητα εκπροσωπώντας την υπηρεσία που εκπροσωπώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Δεν νομίζω ότι έχω περισσότερες πληροφορίες από αυτές που έχετε εσείς κυρία ε, Γκόμες σχετικά με την στήριξη προς τον κύριο Μπραήμι. Λοιπόν, έχουμε πει επανειλημμένα ότι μπορούμε να τον στηρίξουμε. Αν θέλει ε, βοήθεια όσον αφορά την επιμελητία, βοήθεια δηλαδή προς την προσωπία στη Δαμασκό, μπορεί να την έχει. Δεύτερον, εάν χρειάζεται πολιτική βοήθεια, βεβαίως και αυτή μπορεί να κινητοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Και τέλος, η ύπατη εκπρόσωπος θέλει να συνεργαστεί μαζί του έτσι ώστε να έχουν κάποιες κοινέ απόψεις όσον αφορά την ενδεχόμενη επίλυση ε, της, ε, ε, του προβλήματος. Άλλωστε θα το συναντήσει την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Τώρα, ξέρετε ότι στον ε, ε, διάλογο για τα πυρηνικά έχουμε συχνό διάλογο και πρόσφατο μάλιστα με τον κύριο Τζαλίλη. Στη διάρκεια των επαφών μπορεί να μιλήσουν και για κάτι άλλο εκτός από τα πυρηνικά. για το Ιράν βεβαίως μιλούσαμε προηγουμένως. Όσον αφορά τώρα ε, την επόμενη εβδομάδα ξέρετε ότι θα έχει μια συνάντηση με τον Ζεμπαρή, ο οποίος έχει στενή επαφή με το, με το Ιράν. Επίσης συναντήσαμε ε, τον πρόεδρο Μορσή την προηγούμενη εβδομάδα και γνωρίζετε ότι και ο πρόεδρος της Αιγύπτου και ο υπουργός του των εξωτερικών έχουν πολλές επαφές με το Ιράν. Αναμφισβήτητα λοιπόν η ύπατη εκπρόσωπος δίνει, στέλνει μηνύματα προς το Ιράν ε, ε, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε το Ιράν να συμμετάσχει στην επίλυση του προβλήματος της Συρίας όσον αφορά το Συμβούλιο Ασφαλείας Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενδεχομένως ε, ε, το, το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, κάποια στιγμή θα μπορούσε να φτάσει σε συμφωνία για θέματα όπως αυτό του Συριακού ζητήματος, αλλά ε, τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να, να πω τίποτα άλλο, ακόμα και αν είχα την καλύτερη δυνατή βούληση δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Ε, όσον αφορά το ερώτημά σας για το σεβασμό των συνθήκων της Γενέβης και το κατά πόσον γίνονται σεβαστοί, όχι βεβαίως δεν υπάρχει σεβασμός των συνθήκων της Γενέβης. Το έχουμε πει επανειλημμένα και σας είπα και προηγουμένως ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι στη Συρία έχουμε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας Είπα προηγουμένως ότι η αντιπολίτευση και αυτή δεν έχει τελείως καθαρά χέρια, αλλά δεν είχα καθόλου την πρόθεση και δεν είπα ότι η αντιπολίτευση μπαίνει στο ίδιο επίπεδο με την ε, κυβέρνηση. Βεβαίως το καθεστώς Ασάντ είναι αυτό που έχει κυρίαρχα αίμα στα χέρια του, αλλά ε, ε, τι να σας πω, γίνεται λόγος για βασανιστήρια, γίνεται λόγος για κακή μεταχείριση των αντιφρονούντων. Πρέπει να, το πούμε υπάρχει σεβασμός των συνθήκων της Γενέβης. Όχι, βεβαίως όχι. Τώρα το, ζήτημα είναι ε, διαφορετικό, ε, ε, δηλαδή δεν ξέρουμε εάν θα παρουσιαστεί ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ατιμορρησία. Και όταν είπα ότι εκπρόσωπος μιλάει με τον Υπουργό Λαυρόφ, βεβαίως αναφέρεται στο γεγονός ότι είναι κρίμα, είναι, είναι πρόβλημα που δεν υπάρχει λύση σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργείου Ασφαλείας και το ίδιο αναφέρει και με τον πρέσβη της Κίνας στις Βρυξέλλες. Τώρα, Υπάρχει ακόμα δυνατότητα διαπραγματεύσιμης λύσης, ναι ή όχι. Μερικοί λένε ότι ο Ασάντα έχει πάει πολύ μακριά, έχει προχωρήσει υπερβολικά και επομένως δεν είναι δυνατή πλέον λύση. Είναι πολύ αργά. Αλλά αν είναι πολύ αργά τι έχουμε πια, τι μένει. Η ε, στρατιωτικοί αναλυτές ε, λένε ότι η αντιπολίτευση ε, βράχει πρόθεσμα, δεν είναι σε θέση να κερδίσει. Όλοι οι στρατιωτικοί αναλυτές το λένε. Τώρα, μια εξωτερική ε, ε, στρατιωτική παρέμβαση δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι καθόλου πιθανή, δεν υπάρχει νομική βάση γι' αυτό. Και επομένω, εάν δεν έχουμε δυνατότητα εξωτερική στρατιωτική παρέμβαση, εάν ε, δεν μπορεί να κερδίσει η αντιπολίτευση, επομένω τι μα μένει θα διαπραγματευτούμε μέχρι ότου το επίπεδο του αίματος να φτάσει και να ξεπεράσει το ύψος μας, τι πρέπει να κάνουμε. Ε, δεν υπάρχει βραχυπρόθεσμη λύση, άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να οδεύσουμε προς την, ε, ε, προς την διαπραγμάτευση, προς την πολιτική λύση μέσω της διαπραγμάτευσης. Και εάν μπορέσουμε, αν θέλουμε να πιέσουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας έτσι ώστε να μας δώσει νομική βάση για κάποια άλλη μορφή παρέμβασης, ωραία, ας το κάνουμε. Στρατιωτική βοήθεια προς τη Συρία. Τι να σας πω, δεν είμαι ε, εμπειρογνώμων περί τα στρατιωτικά ε, και δεν έχουμε κι εμείς στην υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση. Μερικοί μεταξύ ημών με ύψιλον ίσως έχετε καλύτερη πληροφόρηση από εμά, αλλά εν πάση περιπτώσει εάν δεν υπήρχε βοήθεια εξωτερική νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είχε κρατήσει ο Άσαντ μέχρι τώρα λέτε ε, πόσο κίνδυνος υπάρχει να, η επόμενη μέρα να είναι στη Συρία όπως στη Λιβύη ή σε άλλες χώρες. Ε, τι να σας πω, εγώ νομίζω ότι ε, η τελική, ο τελικός απολογισμός της Αραβικής Άνοιξης πρέπει να έχει περισσότερες αποχρώσεις από αυτό που αναφέρατε εσείς. Δηλαδή, ωραία λέω, λέμε ότι τα πράγματα δεν είναι εξαιρετικά, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι στη Λιβύη κατάφεραν πρώτον να ξεφορτωθούν ένα τύρανο, να έχουν μεταβατική περίοδο, να κάνουν εκλογές, ε, να έχουν κυβέρνηση βάσει εκλογών οι οποίες εκρίθησαν αξιοπρεπείς, κυρίως για χώρα η οποία επί σειρά δεκαετιών είχε δικτατορία και επομένως η εκτίμηση που κάνουμε εμείς, η αξιολόγηση που κάνουμε εμείς ε, για την Τινησία, για τη Λιβύη, για την Αίγυπτο, για την Αραβική Άνοιξη είναι λίγο πιο, έχει περισσότερες αποχρώσεις. Ε, δεν λέμε ότι όλα είναι ρόλο ότι όλα είναι καλά, αλλά καταλαβαίνετε ότι μετά από τόσα χρόνια θεοκρατικών καθεστώτων ή αυταρχικών καθεστώτων όλα δεν μπορεί να κυλήσουν ε, πάνω σε μετάξι, αλλά βεβαίως ε, ε, πολλά πράγματα έχουν γίνει καλά και αν μπορούσε η Συρία να έχει μία αντίστοιχη εξέλιξη δεν θα ήταν και τόσο κακό. Κυρία Μπλονέρα εάν ένα μέρος της ε, ε, ανθρωπιστικής βοήθειας ε, το, του Ερυθρού Σταυρού δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά, τι να σας πω, πρώτη φορά το ακούω αυτό, θα μιλήσω και με τους συναδέλφους της ΕΚΟ, της ανθρωπιστικής βοήθειας και αν έχετε εσείς επιπλέον πληροφορίες παρακαλώ να μου τις δώσετε και να τις δώσω και εγώ με τη σειρά μου στους συναδέλφους ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά πρώτη φορά ακούω κάτι τέτοιο. Όμω δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω. Δεν μπορώ να διαψεύσω, αλλά δεν μπορώ και να επιβεβαιώσω. Εάν έχετε πληροφορίες, παρακαλώ να τις δώσετε για να τις ε, διαβιβάσετε στους συναδέλφους της ΕΚΟ και θα το κοιτάξουν το θέμα από κοντά. Η δεύτερη ερώτησή σα, ε, ε, ε, ερώτηση που δεν θα ήθελα να ε, μου θέσετε, εάν θα ζητήσουμε τους Ισραηλούς να ανοίξουν τα σύνορα, τι να σας πω. Βαθύς αναστεναγμός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι το να, ζητήσουμε, ε, να τους ζητήσουμε να ανοίξουν τα σύνορά τους προς τη Συρία ίσως ε, φαντάζομαι ότι δεν θα τους αρέσει πάρα πολύ. Ίσως θα μπορούσε να θέσει κάποια προβλήματα αυτό στην ε, ασφάλεια. Τώρα, εάν ε, ε, ε, έχουμε περιθώριο να υποβάλουμε το ερώτημα, το βέβαιο είναι ότι θα διαβιβάσω το ερώτημα στην, στους πολιτικούς μου προϊσταμένους και βεβαίως πραγματικά, όχι, δεν θα το πω στο στήλο ότι η κυρία Μπρόνα δεν θέλει να το σκεφτείτε, το, θα το πω με μεγάλη σοβαρότητα. Όσον αφορά τώρα την no-fly zone, Ξέρετε ότι ε, ε, εάν ε, ε, θέλουμε να έχουμε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο ή μια buffer zone. Αυτό, αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ε, με την στήριξη της ε, Συρίας γιατί διαφορετικά και δεν θέλω εδώ να μιλάμε μόνο έτσι δικολαβίστικα και βάσει των διεθνών συνθήκων για να κρυβόμαστε πίσω από αυτές. Υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο. Ξέρετε ότι δεν μπορούμε εύκολα να έχουμε ένα ψήφισμα που να επιτρέπει στη διεθνή κοινότητα ε, να διασφαλίσει μονάχα έναν ανθρωπιστικό διάδρομο στην ε, Συρία. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε την Κίνα, έχουμε την Ρωσία. Δεν θα είναι εύκολο να ε, περάσουν τέτοιες αποφάσεις, αλλά βεβαίως από την άλλη πλευρά, μια και κάθε μέρα έχουμε σφαγές αμάχων, κάθε μέρα χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τα προσκόμματα. Ευχαριστώ πολύ. Your Excellency. Ευχαριστώ. Εξοχότατε κύριε Πρέσβη. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο πιο γρήγορα μπορώ σε ερωτήσεις. Ξέρω ότι ο χρόνος σας τελειώνει. Ο κύριος Μιγκαρέλη ε, απάντησε εκτενέστατα. Ε, εσείς ρωτήσατε για τη στρατιωτική επιλογή και την ε, ζώνη απαγόρευση υπέκτηση και τι μπορούν να κάνουν χώρες. Τα στρατιωτικά και no-fly zone, όλα αυτά έχουν συζητηθεί και όλοι φρονούν, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι φρονούν ότι είναι μια καλή πίεση η No-Fly Zone. Ο Υπουργός Εξωτερικών πριν από λίγες εβδομάδες ήταν στη Νέα Υόρκη και δήλωσε και αυτό ότι θα πρέπει να βρούμε κάποιο ε, τρόπο να τα σταματήσουμε αυτά. Αλλά όπως γνωρίζετε το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, το απέτρεψε. Μόνοι μας οι μερικές χώρες δεν γίνεται αυτό, είναι ανέφικτο και αδιανόητο. Θα πρέπει να είναι απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας η επιβολή κυρώσεων. Μέχρι να γίνει αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα καμιά στρατιωτικής επέμβασης. Και αν το κάνει μία χώρα θα υποστεί επικρίσεις. Μπορεί στην αρχή να τη χειροκροτήσουν αλλά μετά θα τη λιθοβολήσουν. ό,τι αφορά το ΠΚΚ και τα ζητήματα εκεί, εξεπλάγει από την ερώτηση του κυρίου Χαζηγεωργίου για αυτό το θέμα. Η κατάσταση στη Συρία και την Τουρκία δεν συγκρίνεται. Δεν μπορούν να συγκριθούν τα δύο. Εδώ μιλούμε για ένα καθεστώς που δεν επέτρεψε καμία ε, ε, αντιπολίτευση που την καταπνίγει και ακριβώς ε, επειδή δεν υπήρχε ποτέ αντιπολίτευση, ήταν πάντα απαγορευμένη, έχουμε αυτό το φαινόμενο. Από την άλλη έχουμε μια χώρα δημοκρατική. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Τι διαπιστώνουμε. Οι δραστηριότητε του ΠΚΚ δεν είναι ε, τυχαίε. Έχει αναγνωριστεί ως τρομοκρατική ε, οργάνωση από τους 27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εκπροσωπεί τους Τούρκους. Είναι τρομοκρατική οργάνωση. Γι' αυτό ε, ευχαριστώ τα επιχειρήματα του κυρίου ε, Σαλαφράνκα που είπε ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η Τουρκία στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Για τους συνοριακούς ελέγχους. Ναι, κάποιους ε, μεθοριακούς σταθμούς από την άλλη πλευρά τους ελέγχει αντιπολίτευση. Και έχουμε δει ότι ορισμένοι ελέγχονται ακόμα από την κυβέρνηση, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως σας είπα, από την αντιπολίτευση. Και επιτρέπουμε στους Σύρους να έρχονται ε, στην Τουρκία, γιατί ευτυχώς ε, έχουμε σύστημα ε, που δεν χρειάζεται θεώρηση διαβατηρίων. Είναι πολύ εύκολο να μπουν στη χώρα. Ναι, βεβαίω μοιάζει όλο και περισσότερο με εμφύλια σύραξη και έτσι θα πρέπει να αποκαλείται. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονό ότι παρόλα αυτά δεν μπορούμε να επέμβουμε, όπω και να το ονομάσουμε. Το είπε και ο κύριο Μιγκαρέλη ξεκάθαρα υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί κανείς να επέμβει στη χώρα αυτή. Πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Υποθέτω ότι θα πρέπει να ε, αφαιθούμε στην αντιπολίτευση ε, η οποία θα πρέπει να συνέλθει, να οργανωθεί. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε όπλα, παρά μόνο ανθρωπιστική βοήθεια, να τους οργανώσουμε, να τους ε, κάνουμε πιο αντιπροσωπευτικούς, να συμπεριλαμβάνουν και περισσότερες απόψεις, ε, αλλά τα πράγματα πριν βελτιωθούν θα χρειαστεί να ε, ε, Κάποιες χώρες μπλοκάρουν ακόμα την οποιαδήποτε δράση και βλέπουμε ότι ε, χάνεται ο έλεγχος, ξεφεύγει η κατάσταση. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες ε, για να πείσουμε εκείνους που είναι ακόμα διστακτικοί ότι είναι η ώρα να δράσουμε, αλλιώς θα είμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Θυμηθείτε τι έγινε στη Βοσνία, στην Αφρική και αλλού. Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε και αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Δυστυχώς έτσι έχει πραγματικότητα αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Δεν ξέρω, ξέχασα καμία ερώτηση. Νομίζω ότι απάντησε τις περισσότερες ο κύριος Μιγκαρέλη. Αν υπάρχουν και άλλες που ξέχασα, παρακαλώ να μου το πείτε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μιγκαρέλη, ευχαριστώ εξοχότατε ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ανταλλαγή απόψεων θα γίνει με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαλή, άτυπη εδώ σε λίγα λεπτά, χωρίς δερμηνία.